Σας λέει η πρόεδρος. Γεια σας σε όλους. Πού είναι το σφυράκι, λέει. Γεια σας και πάλι. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε για να αρχίσει η συνεδρίαση. Since you have a full house, would you please keep... Είναι γεμάτη η αίθουσα, οπότε κάντε λίγο ησυχία. So, ladies and gentlemen, welcome to all of you. Καλώς ορίσατε όλοι κυρίες και κύριοι. Πρώτα-πρώτα καλώς όρισε η κυρία Μαργκέτ Βεστάγκερ, η οποία ανάλογα με το αποτέλεσμα, το θετικό αν είναι αυτή τη ακρόαση, θα γίνει η εκτελεστική αντιπρόεδρο για την ψηφιακή εποχή. Ε, καλώ όλοι σήμερα στην αίθουσα και όλοι όσοι μα παρακολουθούν στο ίντερνετ. Αυτή η ακρόαση ε, είναι κοινή εκδήλωση τη Επιτροπή Εσωτερική και Προστασία του Καταναλωτή, ΙΜΚΟ, και καλώ ορίσατε, κύριε Ντεσούτερ, και επίση τη ε, Οικονομική Επιτροπή, ΕΚΟΝ. Κυρία Τινάλη, καλώς ορίσατε, πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής, θα συμπροεδρεύσουμε την ε, ακρόαση αυτή. Επίσης καλωσόρισαν τα μέλη της ε, Νομικής Επιτροπής που είναι στην ομάδα για την ακρόαση και της Επιτροπής Απασχόλησης, αλλά άρα και της, και, και Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Η νεοριστής απρόεδρος της Επιτροπής σας ε, εμπιστεύτηκε το χαρτοφυλάκιο της ψηφιακής εποχής, ε, κάτι το οποίο βοηθά τη βιομηχανία και την καινοτομία. Αυτό θα είναι κλειδί για να αναβαθμιστεί η ηγετική θέση της Ευρώπης προς τεχνολογίας αλλά και στρατηγική αυτονομία μας. Ε, επίσης θα ε, είστε επικεφαλής προσπάθειας για μια μακρόπνευση στρατηγία το μέλλον της βιομηχανίας και στρατηγικής για τις ΜΜΕ. Επίσης ε, θα συντονίσετε μια προσέγγιση για την ε, ε, τεχνητή νοημοσύνη και αυτό θα παρουσιαστεί ως έργο για τις πρώτες 100 μέρες της Νέας Επιτροπής και είναι για την Επιτροπή Βιομηχανίας, την Επιτροπή Ήτρε, όλα αυτά είναι βασική μας αρμοδιότητα και γι' αυτό είμαστε μαζί σας κύριε Βέσταγκερ για να ακούσουμε με μεγάλη προσοχή τι έχετε να μας πείτε και έτσι να πετύχει από πλευράς βιομηχανία το έργο σας σε αυτό το χαρτοφυλάκιο και τώρα. Κυρία Ντεσούτερ, έχετε το λόγο. Και τις τρεις μας πρέπει να ακούσετε, λέει η κυρία Ντεσούτερ, Από πλευράς της ε, Επιτροπής ε, ΙΜΚΟ Καλώς ορίσατε, Αντιπρόεδρε Βεστάγκερ, ε, για αυτήν την ακρόαση. Η δική μας Επιτροπή ε, έχει ως αρμοδιότητα τον συντονισμό της εσωτερικής αγοράς, της ενιαίας αγοράς και της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Η ψηφιοποίηση αλλάζει την οικονομία σε κάθε κλάδο της και έχει συνέπειες για επιχειρήσεις, καταναλωτές και όλη την κοινωνία. Είναι από τα μεγαλύτερά μας επιτεύγματα και θα πρέπει τη σημερινή εποχή της ψηφικής αλλαγής να συνεχίσει να αποτελεί μεγάλη μας επιτυχία και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε οι κανόνες της τουρκικής αγοράς να ε, είναι αυτή που πρέπει για την ψηφιακή εποχή ούτω ώστε να έχουμε εμπιστοσύνη του καταναλωτή και να έχουμε ε, καθεστώς θεμητού ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις. Άρα θα πρέπει όλοι να βγουν κερδισμένοι από αυτήν την αλλαγή ισχυρή εσωτερική αγορά σημαίνει να μην έχουμε κατάτμιση, σημαίνει να αποφύγουμε τους τεχνητού διαχωρισμούς μεταξύ ε, των παραδοσιακών αγορών offline και των νέων ψηφιακών αγορών που τους λέμε online. Και η αγορά είναι μία. Διαδικαστικά τώρα θα σας πω ότι σύμφωνα με τις γραμμές για την έγκρισή σας ε, αξιολογούμε τον υποψήφιο επίτοπο τη βάση των γενικών του ικανοτήτων, ε, της ευρωπαϊκής του προσήλωσης και της προσωπικής του εξαρτησίας. Επίσης ε, ζυγίζουμε το πόσο γνωρίζουν το χαρτοφυλάκιό τους και αξιολογούμε και το επικοινωνιακό τους χάρισμα. Πριν από αυτήν την ακρόαση ετοιμάσατε εκείνο το ερωτηματολόγιο, απαντήσατε, όλοι έχουν λάβει τις απαντήσεις και από την Νομική Επιτροπή δεν προβλήθηκε κάποια ένσταση για αυτήν την ακρόαση. Οπότε τώρα θα δώσουμε τον λόγο στην κυρία Τινάλη για την Οικονομική Επιτροπή. Does it work? Οικονομικής Επιτροπής και εγώ σας απευθύνω ένα καλωσόρισμα. Σε όλους που είναι εδώ αλλά κυρίως την κυρία Βεστάγκερ, την γνωρίζουμε καλά στην ε, Επιτροπή μας, ε, διότι είχε το χαρτοφυλάκιο τον αναγνωρισμού κατά την προηγουμένη θητεία ορίστηκε ως που ε, υπεύθυνη για να συνεχίσει το, το έργο της, της Επιτροπής σε αυτήν την ιδιότητα τώρα και τώρα θα είναι η Αντιπρόεδρος για την ψηφιακή εποχή και επίσης θα αναλάβει τον συντονισμό για την ψηφιακή φορολογία και μέχρι τέλος του 2020 θα αναζητήσει την συνένεση σε διεθνές επίπεδο. Η εναλλακτικά θα προταθεί ένας δίκαιος ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος. Σύμφωνα με την προβλόμενη διαδικασία και ο ανταγωνισμός αλλά και η φορολογία είναι βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Σα υπενθυμίζω τα εξή από πλευρά διαδικασία. Πώ θα γίνει αυτή η ακρόαση, θα κάνει εναρκτήρια, αρχική δήλωση κ. Βεστάγκερ μέχρι 15 λεπτά. Επίση, στο τέλο τη ακρόαση θα έχει ένα λεπτό για να κάνει την τελική δήλωση και θα ακολουθήσουν τις εισήγησεις κ. Βεστάγκερ 25 ερωτήσεις από τους ε, βουλευτές. 5 λεπτά ο κάθε βουλευτής και ένα λεπτό ε, συγγνώμη, πέντε λεπτά η κάθε ερώτηση, αλλά θα έχει ένα λεπτό μετά και άλλα δύο λεπτά για απάντηση. Επερωτήσεις επίσης ε, με ένα λεπτό και ένα λεπτό απάντηση. Έχουμε τον πρώτο γύρο των επτά ερωτήσεων των ε, εκπροσώπων των ε, πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων. Επίσης, σας πενθυμίζω ότι θα είμαστε και οι τρεις συμπρόεδροι, πάρα πολύ με τον προβλεπόμενο χρόνο και ουδής θα υπερβεί το προσλεγομενο χρονικο χρονικό όριο. Εάν είναι πάνω από ένα-δύο λεπτά και ερώτηση, δεν θα επιτραπεί η υπερώτηση. Έρχεται σε 23 γλώσσες ε, διερμηνία, οπότε μου μιλήσετε στη μητρική σας γλώσσα, αλλά ε, να έχετε στο μυαλό σας τους διερμηνείς και άρα μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Κύριε έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριες ε, πρόεδροι κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές. Πριν από πέντε χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με επικύρωσε ως ε, Επίτροπο για τον Ανταγωνισμό. Μία πολύ περήφανη στιγμή στη ζωή μου. Μου δόθηκε ευκαιρία να δουλέψω για τους Ευρωπαίους πολίτες σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο για τις αξίες που με καθοδηγούν εδώ και 30 χρόνια. Πάντα ήμουν υπέρ μιας δίκαιης κοινωνίας, όπου ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του, να ακολουθήσει τα όνειρά του, σεβόμενος τους άλλους. Εάν με ορίσετε, θα συνεχίσω να κάνω το ίδιο ως εκτελεστική αντιπρόεδρος για να γίνει η Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή. Πιστεύω ότι θα επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους ε, συνεργαζόμενοι. Αυτό πίστευα όταν μπήκα για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο ως εκπαιδευόμενη. Έκτοτε έχω δει το τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία για να οικοδομήσει μια κοινωνία η οποία ε, λειτουργεί και εκπροσωπεί τους λαούς της και η Ευρώπη θα προσπαθήσει να κάνει περισσότερα. Χαίρομαι για το ότι έχουμε την πρώτη Κομισιόν με ισορροπία φύλων. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις. Να αναφέρω κάποιε. Η κλιματική αλλαγή και ο ψηφιακό μετασχηματισμό θα επηρεάσουν κάθε κομμάτι της ζωή μα. Και καθώ εντείνεται ο παγκόσμιο ανταγωνισμό, θα πρέπει να εργαστούμε σκληρότερα για να υπάρχει ναι, υπάρχουν ίσοι όρια ανταγωνισμού. Έχουμε τα όσα χρειάζονται για να ανταποκριθούμε σε αυτέ τι προκλήσει, εάν συνεργαστούμε. Έχουμε αξίε για τι οποίε μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Ελευθερία, δικαιοσύνη, δημοκρατία. Όλα αυτά έχουν κάνει την Ευρώπη το καλύτερο μέρο για να ζει κανεί. Η Ευρώπη έχει πολλού ανθρώπου με υψηλά προσόντα, εξαιρετικέ υποδομέ δίκαιους και αποτελεσματικούς νόμους. Η ενιαία αγορά δίνει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χώρο για να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να είναι καλύτερες σε αυτό το οποίο κάνουν στον κόσμο. Οπότε, η δική μου δέσμευση δεν είναι να κάνω την Ευρώπη σαν την Κίνα ή την Αμερική. <laughs> Δεσμεύομαι να κάνω την Ευρώπη πιο Ευρώπη. Να οικοδομήσουμε πάνω στα δικά μας δυνατά σημεία και αξίες, έτσι ώστε η κοινωνία μας να είναι ισχυρή και δίκαιη για όλους τους Ευρωπαίους. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχω δει πως η επιβολή των κανόνων του ανταγωνισμού μπορεί να κάνει τις αγορές να λειτουργούν για τους ανθρώπους και όχι αντιστρόφως. Και είμαι υπερήφανη για τη δουλειά που έχουμε κάνει. Υπάρχουν όμως πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Γι' αυτό με τιμά το ότι η πρόεδρος μου ζήτησε να συνεχίσω τη δουλειά μου στο πεδίο του ανταγωνισμού. Θα συνεχίσω να το κάνω με την ίδια ενέργεια και αφοσίωση όπως πάντα. Και με την ίδια προσήλωση στην ανεξαρτησία και την αμεροληψία. Όπως έκανα και πριν από πέντε χρόνια. Γιατί η ανεξαρτησία στον τομέα της επιβολής του νόμου είναι κάτι το αδιαπραγμάτευτο. Οι κανόνες του ανταγωνισμού δεν καθιστούν αξιόπινο το να είναι κανείς μεγάλη εταιρεία. Αλλά οι κυρίαρχε εταιρείε έχουν μια ιδιαίτερη ευθύνη για να μην χρησιμοποιούν αυτή τη δύναμη για να βλάπτουν τους καταναλωτές. Επίσης, οι εταιρείε έχουν δικαίωμα να συγχωνεύονται αρκεί να μπορεί κανείς να τις αντιμετωπίσει. Γιατί οι εταιρείε δεν μπορούν να αρνούνται στου καταναλωτέ τα ωφέλη του ανταγωνισμού τις φθηνές τιμές, την επιλογή των προϊόντων και καινοτόμο προϊόντα που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. Και προφανώς πρέπει να φροντίσουμε και οι κρατικές ενισχύσεις να μην βλάπτουν τον ανταγωνισμό. Γιατί οι Ευρωπαίοι αξίζουν μια οικονομία όπου οι εταιρείε θα ανταγωνίζονται για να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες, όχι απλά να λαμβάνουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις από το κράτος. Είναι δύσκολη καιρή και για τα θέματα του ανταγωνισμού, γιατί οι αγορές αλλάζουν γρήγορα και έχουμε ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές που έρχονται. Αλλά η ανθρώπινη φύση, τα βασικά κίνητρα, όπως ε, ο φόβος και η απληστία, δεν αλλάζουν. Οπότε, οι αρχές οι οποίες μας καθοδηγούν έχουν την ίδια σημασία σήμερα όσοι είχαν και πριν από 60 χρόνια όταν υπογράφηκε η συνθήκη της Ρώμης. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε ο τρόπος εφαρμογής αυτών των αρχών να ταιριάζει σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα. Οπότε, θα ξεκινήσω με την εξέταση των κανόνων περί αντιτράστ, συγχωνεύσεων και κρατικών ενισχύσεων. Και στη διαδικασία αυτή θα μας βοηθήσουν τα όσα μάθαμε εξετάζοντας το πώς η ψηφιοποίηση επηρεάζει τον ανταγωνισμό, μεταξύ των οποίων και η έκθεση των τριών ειδικών συμβούλων. Θεωρώ ότι ο δίκαιος ανταγωνισμός είναι σημαντικός για να προετοιμάσει την οικονομία μας για τις προκλήσεις που έρχονται. Αλλά ο ανταγωνισμός δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική για το βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης, που θα βασίζεται σε αυτά τα οποία καθιστούν την Ευρώπη ανοιχτή. Στο ότι είναι ανοιχτή και ποικιλόμορφη. Οπότε η βιομηχανική στρατηγική πρέπει να είναι για όλους. Πρέπει να είναι πράσινη και πρέπει να βασίζεται στον δίκαιο ανταγωνισμό. Και βεβαίως αυτό θα περιλάβει και την χάραξη μιας νέας στρατηγικής για την καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις μικρές και μεσαίες εταιρείες. Μαζί συναποτελούν πάνω από το μισό του εισοδήματο των επιχειρήσεων της Ευρώπης, δύο τρίτα των εργαζομένων και παρέχουν την κατάρτιση που χρειάζονται οι νέοι μας. Και, βασικό, αυτό το οποίο ζητάνε από εμά είναι να δημιουργήσουμε μια δίκαιη αγορά και να μην υπάρχουν τα εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους. Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει επίσης να συνεργαστούν. Αυτό σημαίνει μια πιο στρατηγική χρήση των δημοσίων προμηθειών, περισσότερη χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία. Και αυτό σημαίνει συνεργασία με τα κράτη-μέλη σε σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Θα έχουμε ολόκληρες αυτές τις αλυσίδες αξίας από τα πανεπιστήμια, στους προμηθευτέ, τους κατασκευαστές, μέχρι αυτούς που ανακυκλώνουν τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία. Και η στρατηγική αυτή πρέπει να πάει πέρα από την ενιαία αγορά. Καθώς γινόμαστε όλο και πιο αλληλένδετοι, επηρεαζόμαστε όλο και περισσότερο από τις αποφάσεις που λαμβάνουν άλλοι. Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο 80 χωρών, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Οπότε είμαστε σε μια ισχυρή θέση για να επιβάλλουμε παγκόσμιου όρου ανταγωνισμού. Αυτό περιλαμβάνει τι προτάσει μα για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε οι ξένες κρατικές επενδύσεις και επιδοτήσεις να μην υπονομεύουν τον δίκαιο ανταγωνισμό. Επίσης, η σωστή βιομηχανική στρατηγική σημαίνει ότι η Ευρώπη θα είναι καλή και έτοιμη για την ε, ψηφιακή εποχή. Υπάρχουν δύο ειδών επιχειρήσει. Αυτέ που είναι ήδη ψηφιακέ και αυτές που θα γίνουν ψηφιακέ. Και η ψηφιοποίηση έχει πάρα πολλέ δυνατότητε για να βελτιώσει τη ζωή μα. αλλά για να τι εκμεταλλευτούμε αυτέ, χρειαζόμαστε του κατάλληλου κανόνες για να έχει ο κόσμος την απαραίτητη εμπιστοσύνη στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πρέπει να σέβεται τους πολίτες ε, και τις θεμελιώδεις αξίες μας. Σήμερα θα ήθελα να τονίσω τρεις βασικές αξίες. Εμπιστοσύνη, ανθρωπιά και δικαιοσύνη. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα για το τι θα κάνω τα επόμενα πέντε χρόνια. Περί εμπιστοσύνης. Πρέπει να δούμε τις ανησυχίες των ανθρώπων για την τεχνολογία και έτσι να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη. Θα εργαστώ σε ένα νομοθέτημα περί ψηφιακών υπηρεσιών το οποίο θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση των κανόνων ευθύνη και ασφαλείας για τις ψηφιακές πλατφόρμες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα. Και χρειάζεται να ρυθμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείε συλλέγουν και μοιράζονται δεδομένα, έτσι ώστε να ωφεληθεί ολόκληρη η κοινωνία. Επί της ανθρωπιάς. Χρειαζόμαστε κανόνες έτσι ώστε να χρησιμοποιείται δεοντολογικά η ε, τεχνητή νοημοσύνη. Να μην υπονομεύει τις ανθρώπινες αποφάσεις. Θα υποβάλω λοιπόν κάποιες προτάσεις για την ευρωπαϊκή προσέγγιση στην ε, τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια των πρώτων 100 ημερών και για την δικαιοσύνη. Οι δίκαιε συνθήκες εργασία και φορολογία είναι τα θεμέλια μιας σωστή κοινωνίας, οπότε πρέπει να φροντίσουμε όσοι εργάζονται σε πλατφόρμες να έχουν σωστέ συνθήκε εργασία και ότι οι ψηφιακές εταιρείε θα πληρώνουν το φόρο που του αναλογεί. Θέλουμε οι κανόνε αυτοί να βασίζονται σε μια παγκόσμια συμφωνία και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, μέχρι το τέλος του 2020 θα αναλάβουμε δράση. Οπότε, έχουμε προκλήσεις μπροστά μας. Όχι μόνο να ορίσουμε, αλλά και να εφαρμόσουμε τους κατάλληλους κανόνες, έτσι ώστε οι αγορές να σέβονται τις θεμελιώδεις αξίες μας και να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης που θα κάνουν τις ζωές μας καλύτερες. Είτε μιλάμε για την υγεία, τις μεταφορές, είτε για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για το σκοπό αυτό. Ελπίζω. Και έχω την πεποίθηση ότι θα συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία πέντε χρόνια. Έχω συζητήσει συχνά προτάσεις και ιδέες με βουλευτές και νομίζω ότι ο πραγματικά ανοιχτό διάλογος ε, κατέσε δυνατή την υιοθέτηση νέας νομοθεσίας. Εάν με ναι. επιβεβαίωστε στην θέση μου, θα συνεχίσω να ε, συνεργάζομαι μαζί σας με τρόπο ανοιχτό, με συνεργασία σε κάθε βήμα της νομοθετικής διαδικασίας και αναμένω και την συνεργασία με τις επιτροπές σας. Εξάλλου, η Ευρώπη είναι ομαδική εργασία και σήμερα που αντιμετωπίζουμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής μας, χρειαζόμαστε πιο πολύ από ποτέ να συνεργαστούμε έστι έτσι ώστε η Ευρώπη να παραμείνει το καλύτερο μέρος για να ζει κανείς. Ειδικά αν είναι κανείς γυναίκα. Thank you. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Βεστάγκερ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Αντρέα Σφάπα από την Επιτροπή ΙΜΚΟ και από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Οριστήσα Επίτροπε, σα καλωσορίζουμε. Ήσασταν κρυφό αστέρι της Επιτροπής Ιούνκερ και ε, χρηματοπιστωτικές ανάγκες ε, σας σε ακόμα μεγαλύτερο αστέρι σήμερα. Συγχαρητήρια. Έχουμε πραγματικές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, ιδίω ε, σε σχέση με το χαρτοφυλάκι που έχετε αναλάβει εσείς. Η ψηφιακή αγορά είναι γεμάτη κρυφά άστρα που όμως δεν λάβουν και τόσο πολύ και θα συνεχίσω στα γερμανικά. Η οικονομία ψηφιακών πλατφορμών σίγουρα παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές. Υπάρχουν όμως ρυθμιστικοί φραγμοί που είναι το σημαντικότερο εμπόδιο για τις επιχειρήσεις αυτές και δεν τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν γρήγορα και όχι μόνο στο ψηφιακό τομέα αλλά και στους κλασικούς βιομηχανικούς τομείς όπου παρατηρείται ε, ε, μία πίεση ε, σε ό,τι αφορά το διεθνή ανταγωνισμό πολλές φορές ε, συνοδεύεται και από οικονομική ενίσχυση και απειλεί τους Ευρωπαίους πρωταγωνιστές. Όλοι οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν από τις συγχωνεύσεις καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερα προϊόντα. Αυτά τα αξιώματα τα ευρωπαϊκά τα υποστηρίζετε και ποια είναι τα μέτρα που προβλέπετε να ακολουθήσετε εσείς και η Κομισιόν υπό τη δική σας καθοδήγηση για να ε, διευκολύνει τα πράγματα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, και να ε, υπάρχουν δυνατότητες ισότιμου ανταγωνισμού απέναντι δύο στην Ανατολή και να διατηρηθούν τα πλονεκτήματα των επιχειρήσεων της Ευρώπης. Ευχαριστώ απάντηση. Πράγματι, πολύ σωστά λέτε ότι εδώ ουσιαστικά έχουμε δύο προκλήσεις, μια διτή πρόκληση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε στην εσωτερική αγορά αφενό τον δίκαιο ανταγωνισμό ε, για να έχουν τα προϊόντα και υπηρεσίες οι καταναλωτές μας. Και επίσης να προστατεύουμε τις δικές μας επιχειρήσεις από τον αθέμητο ξένο ανταγωνισμό. Και δεν το ε, βλέπουμε αυτό μόνο με τη δέστησή μα ή δεν το αντιλαμβανόμαστε μόνο, αλλά έχουμε και απτά στοιχεία. Βλέπουμε, παραδείγματο χάρη, να μην εξασφαλίζεται χρηματοδότηση με τον ίδιο ανταγωνιστικό τρόπο από τι ξένε επιχειρήσει από για τι ευρωπαϊκέ που ισχύουν αυστηροί κανόνε. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε σημαντικά βήματα και κάναμε κάποια από αυτά. Για παράδειγμα, προτείναμε μία αλλαγή. Παραδείγματο χάρη, σε ό,τι αφορά τι σχέσει μα με την Κίνα που δεν είναι αναψώμενη οικονομία, το κάθε άλλο. Είναι στρατηγικό εταίρο σε κάποιου τομεί όπω η κλιματική αλλαγή, αλλά είναι και στρατηγικό ανταγωνιστή. Και θα πρέπει σε αυτό να αντιδράσουμε. Και εδώ πραγματικά ελπίζω να συνεργαστώ με τους συναδέλφους ώστε να έχουμε τα ε, εργαλεία για τις ε, δημόσιες προμήθειες. Χρειάζεται αμοιβαιότητα και να καλούμε ξένε επιχειρήσει στι δικέ μα αγορέ, αλλά να ισχύει και το αντίστροφο, να μπορούμε και εμεί να έχουμε πρόσβαση στι ε, ξένε αγορέ και μιλάμε για το 15% του ΑΕΠ και με τους ξένους θέλουμε να επενδύουν αλλά για τους σωστούς σκοπούς στην Ευρώπη. Φυσικά και καλωσορίζουμε τους επενδυτές. Θα πρέπει να έρχονται όμως για επιχειρηματικούς σκοπούς. Ένα από τα ανοιχτά θέματα είναι αν μια κρατική επιχείρηση από το εξωτερικό αγοράζει μια επιχείρηση, αλλά έρχεται εδώ ουσιαστικά με ξένη ενίσχυση για να υπονομεύσει ε, τον δίκαιο ανταγωνισμό, θα πρέπει να βρούμε κάποια λειτουργικά εργαλεία για να προστατεύσουμε τι επιχειρήσει μα ε, πάντα στο πλαίσιο τη ίδια αγορά. Δεν τα έχουμε ακόμη, αλλά είναι μεγάλη προτεραιότητα για εμά. 30 δευτερόλεπτα έχετε. Σίγουρα είπατε ότι πρέπει να συνεργαστείτε με το συναδέλφου σας αλλά πρέπει να μας πείτε ε, τι θα γίνει με τα μέτρα, παραδείγματος χάρη των αμερικανικών επιχειρήσεων, με μονομένα ε, τέτοια μέτρα κατά συγκεκριμένων επιχειρήσεων πολλές φορές τα έχουμε ζητήσει. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι και στον ψηφιακό τομέα στο μέλλον θα μπορούν να, να χρησιμοποιηθούν οι κανόνες για το δίκαιο ανταγωνισμό, για να μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Well, this has Πράγματι, σίγουρα εγκράστηκα εντατικά και κάποιες φορές ε, με απογοήτευσαν οι εξέλιξεις πρέπει να σας πω, γιατί σίγουρα ε, πολύ ταχύς, ε, ταχύες είναι οι αλλαγές και σίγουρα είναι δύσκολο, ε, δεν μπορεί κανείς να κάνει τις αρχές επιβολής του νόμου να εργαστούν ακόμα πιο γρήγορα. Αυτό θα έπρεπε να γίνει όμως και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Υπάρχει τώρα αυτή η υπόθεση λέμε σε μια επιχείρηση πρέπει να σταματήσει αυτά που κάνεις γιατί βλάπτεις τον ανταγωνισμό. Και αν σταματήσεις, έπειτα θα προχωρήσουμε με τη διαδικασία για να αποδείξουμε κατά πόσον ναι, έχει υπάρξει ζημία ή όχι. Δηλαδή έχουμε ακολουθήσει μια διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων ε, προς το παρόν. Πάντως είναι προτεραιότητά μας, τον επιταχύνουμε την προσπάθεια στον τομέα αυτό. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Πολ από ΕΚΟΝ, ε, Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κυρία Βεστάγκερ. Συγκέντρωση ε, χρήματος και δύναμης είναι το αρνητικό στοιχείο, αρνητική όψη της ψηφιακής εποχής. Οι φορολογικοί γίγαντε, ε, οι μεγάλε πολυεθνικέ δεν πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρου και αυτό προκαλεί μεγάλε αντιδράσει. Εσεί θα ζητήσετε για ένα φόρο ψηφιακών υπηρεσιών αν δεν δώσουν αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσει σε επίπεδο Συμβουλίου. Θα συνεχίσετε να ε, ασχολείστε με τέτοιε υποθέσει, ε, ενώ ξέρουμε τι έγινε με την υπόθεση Starbucks. Και επίση, έχουμε τεχνολογικού Αμερικανού ε, γίγαντες. Ε, δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι ανταγωνιστές ε, να έχουν ε, δίκαιο ανταγωνισμό με αυτές τις επιχειρήσεις. Τι θα κάνετε για να αλλάξει κατάσταση ριζικά, για να έχουμε ευρωπαϊκή επιτυχία και επίσης τα δεδομένα μας, τα δεδομένα των Ευρωπαίων καταναλωτών και χρηστών να είναι προστατευμένα ώστε να μην μπορούν να τα καταχραστούν οι Αμερικανικοί αυτοί γίγαντες. Uh, Πρώτα απ' όλα, ελπίζω να μας ακούν και τα κράτη-μέλη. Γιατί αυτές ε, οι υποθέσεις με τις κρατικές ενισχύσεις δεν θα μας δώσουν ένα δικαιοφορολογικό σύστημα. Πρέπει να αλλάξει νομοθεσία γι' αυτό. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η εταιρική φορολογία ανακαλύφθηκε πολύ πολύ πριν ε, δει το φως της ημέρας ο πρώτος υπολογιστής. Και η εταιρική φορολογία πρέπει να ψηφιοποιηθεί επίσης. Αλλιώς ε, οι, οι επιχειρήσεις θα συνεισφέρουν όλο και λιγότερο στις ε, κοινωνίες όπου και παρέχουν ε, τις υπηρεσίες τους. Σίγουρα δεν είναι δίκιο κάποιες επιχειρήσεις να αποκομίζουν όφελος μόνο αυτές. Και ε, υπάρχουν οι υποθέσεις που είναι ανοιχτέ. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μας πούν πώς χρησιμοποιούν αυτές τις φορολογικές συμφωνίες, τα λεγόμενα tax rulings όπω κάναμε και πριν από δύο χρόνια περίπου σε μια συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλά για του φόρου, ναι, θα συνεχίσουμε και ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ε, γενική συμφωνία, παγκόσμια συμφωνία, όπω κάναμε ε, για να αποφύγουμε τη μετατόπιση κερδών και τη διάφορη φορολογική ε, βάση. Και είναι τώρα νομοθεσία αυτό. Αν όμω δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, ναι, θα αναλάβουμε μόνοι μα δράση. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να πιέζουμε και τα μεμονωμένα κράτη-μέλη που το κάνουμε γιατί οι επιχειρήσεις ζητούν δίκαιη φορολογία και πρέπει να αποκριθούμε στο αίτημά τους. Είναι προτεραιότητά μας λοιπόν και σε ό,τι αφορά το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν την νομοθεσία, που παρανομούν. Τα πρόστιμα, γιατί είπατε για το Starbucks, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του τζίρου, 4 με πρέπει να δούμε προ το μέλλον. Και το μέλλον ε, δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Πρώτον, πρέπει να του πούμε σταματήστε αυτά που κάνετε. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι που έχει το ίδιο αποτέλεσμα αυτό που κάνετε πριν. Και φυσικά έχουμε στην εργαλειοθήκη μας περισσότερα εργαλεία για να ε, ξαναφέρουμε τον ανταγωνισμό σε αυτή την αγορά. Και σίγουρα θα γινόμαστε όλο και σοφότεροι και θα καταλαβαίνουν και αυτοί καλύτερα τι ε, επιπτώσεις θα έχουν, παραδείγματος χάρη τα λειτουργικά συστήματα, Κίνα κτλ. Υπάρχει υπερώτηση. Ναι, ναι, ε, καλό το ότι ξυπνάμε όλα και περισσότερο, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε τίποτα για να ανασχέσουμε αυτή την εισβολή των ε, γιγάντων της αγοράς. Άρα, εσείς τι νομίζετε ότι έχετε ως αποτελεσματικό όπλο για να καταπολεμήσετε αυτά τα ε, μονοπόλια. Πώς θα γίνει να υπάρξει κάποιος ανταγωνισμός. Το έχει πει αυτό το κοινοβούλιο. Ε, το facebook ή για κάποια άλλη εταιρεία. Κάτι θα πρέπει να γίνει. Ναι, πέρα από το θέμα του λειτουργικού ήταν το θέμα των browsers που θα που ήταν ένα από τα επεισόδια του serial της Google. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει χώρο στην αγορά, αλλιώς με αυτή την παράνομη τακτική καταλαμβάνουν όλο το χώρο αυτές τις εταιρείε. Τώρα όσον αφορά την κατάδυμηση των των μεγάλων εταιρεών αυτό μπορεί να γίνει, έχουμε το εργαλείο, θα πρέπει όμως να δούμε πώς θα είμαστε όσο γίνεται λιγότερο παρεμβατικοί για να υπάρχει υγιή συνταγωνισμό, γιατί ακριβώς δεν είναι και λίγο το να σπάσει σε κομμάτια μια μεγάλη εταιρεία και βέβαια θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το πιο δόκιμο μέσο. Άλλο, και πολλέ φορέ αυτό υποτιμάται, ότι εμεί ω καταναλωτές βλέπουμε τους Αμερικανούς ως γίγαντες αλλά και οι Αμερικανοί το ίδιο για τις ψηφιακές υπηρεσίε τους ε, Ευρωπαίους και στο hardware και για το λογισμικό και μεταξύ επιχειρήσεων ε, η Ευρώπη πολλά μπορεί να καταφέρει. Νίκολα, Μπίερ, Ήτρε, Renew Europe. Ευχαριστώ. Ε, πολύ συναρπαστικό το εγχείρημα να κάνετε την Ευρώπη κατάλληλη την ψηφιακή εποχή. Βλέπω ότι ε, σας απασχολεί και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνητή νοημοσύνη που πολλά υπόσχεται για την ανθρωπότητα στο μέλλον και μπορεί να ωφελήσουν αυτές οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της υγείας, ε, στην ατομική καλύτερη παιδεία, κινητικότητα για άτομα με αναπηρία, ε, βελτίωση του περιβάλλοντος, μεγαλύτερη προστασία για τους πολίτες. Όλα αυτά μπορεί να τα εγγυηθεί για τους πολίτες και για την οικονομία, άρα προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες. Συμφωνείτε μαζί μας ε, ότι το παραγωγικό καινοτόμο δυναμικό της τεχνητής νομοσύνης ε, θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε ε, γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσει ε, και περιορισμοί και θα πρέπει στρατηγικά να κινηθούμε ώστε όχι μόνο να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό αλλά να είμαστε και πρωτοπόροι ε, ως Ευρώπη. Τι μπορούμε λοιπόν να, να περιμένουμε από εσά το επόμενο, την επόμενη πενταετία με καλά παραδείγματα συγκεκριμένα. I Συμφωνώ, λέει κύριε Βεσταγιώνα Συμφωνώ ότι υπάρχει δυνατότητα, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι και όλο είναι και περισσότερο χάνει την πιστοσύνη του κόσμου στην τεχνολογία. Οπότε για να μπορέσουμε να έχουμε τα υπέρ θα πρέπει να ανεβάσουμε την εμπιστοσύνη ότι δηλαδή η τεχνολογία εξυπηρετεί τους πολίτες, εξυπηρετεί τους ανθρώπους και για την τεχνητή νοημοσύνη είχαμε μία ομάδα υψηλού επέδου κατέληξαν σε 7 κατευθυντήριε για το πώ είναι δυνατόν να αυξηθεί η εμπιστοσύνη προς την τεχνητή νοημοσύνη και αυτό δεν είναι σκίση επί χάρτου. Αυτό είναι κάτι που στην πράξη οφείλει τι επιχειρήσει, διότι πάρα πολλέ ε, επιχειρήσει ε, συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τι κατευθυντήριε ε, όταν χρησιμοποιούν τέλο πάντων την τεχνητή νοημοσύνη το Δεκέμβριο. Οπότε επενδύουμε και Πρέπει να δώσουμε καταλαβή ο κόσμο ότι εδώ. Μπορεί να λέμε ότι τα έχουν όλα οι Κινέζοι, τα δεδομένα και οι Αμερικανοί όλα τα λεφτά, αλλά εμείς εδώ έχουμε στόχους. Και η τεχνητή νοημοσύνη εδώ στην Ευρώπη ωφελεί στο περιβάλλον, στην υγεία, στις ε, μεταφορές. Ακριβώ εκεί θέλουμε η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιηθεί για έναν πιο σπουδαίο σκοπό Άρα χρειάζεται η έμπνευση για να δούμε τι θα γίνει με τα δεδομένα, πού θα ξεβρεθούν οι πόροι, πώ θα επενδύσουν περισσότερο, γιατί φυσικά και χρειάζονται περισσοτερε επενδύσεις. Ε, τρεις ή τέσσερις φορές λιγότερο επενδύουμε από του άλλου. Καλά τα δεδομένα, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι θέλουμε να πετύχουμε και αυτό θα είναι το κίνητρο. Η πρόεδρο και τώρα η Αλεξάνδρα Α, όχι, όχι, συγγνώμη, ξέχασα ότι έχετε και ερώτηση. Ναι, σύντομα. Πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να επενδύσουμε σε αυτέ τι τεχνολογίε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό ταυτόχρονα, όπω να υπερασπιστούμε τι αξίε μα. Τα επόμενα πέντε χρόνια πώ θα πετύχετε από κοινού μαζί με τα κράτη-μέλη να μπορέσουμε να ε, έχουμε μια συγκέντρωση και κοινή αξιοποίηση όλων αυτών των δυνατοτήτων και να μην ε, υπάρξει κατακαιρματισμός. Πρώτα πρώτα, ο προϋπολογισμός για την επόμενη επταετία να εγκριθεί και έτσι να σταθούμε στη δουλειά. Και η Επιτροπή μας πρότεινε να αυξηθούν οι επενδύσεις αρκετά, ούτως ώστε να μπορέσουμε όλα αυτά να τα καταφέρουμε. Δεύτερον, έχουμε πιο στατική χρήση των ε, ε, προμηθειών και των δημοσίων συμβάσεων Πάρα πάρα πολλά. Μιλάμε για ξαψήφια ποσά που δίνουμε. Άρα θα πρέπει να πιστούν και οι μικρότερες επιχειρήσεις ότι μπορούν να τα καταφέρουν και έτσι να έχουμε μια στρατηγική τέχνη της νοημοσύνης για περισσότερους τομείς της κοινωνίας. Έχουμε τώρα κάποιους κόμβους καινοτομίας και Έχουμε νεοφύης επιχειρήσεις σε πολλούς τομείς και άρα νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε πρόεδρος. Αλεξάνδρα Τζίζ, ΙΜΚΟ για τους πράσινους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Αντιπρόεδρε, η οδηγία της επιχειρήσης θα ωφελήσει, μιλάμε για μεγάλο ποσό του έπαρα, επίσης οι πολίτες και οι καταναλωτές έχουν σήμερα πρόβλημα. Έχουμε, έχουμε παραπληροφόρηση, έχουμε παρεμβάσεις στον τομέα της πολιτικής, όλα αυτά επηρεάζουν τους καταναλωτές. Έχουμε αυτόν τον καπιταλισμό της επιτήρησης. Θέλω να υποσχεθείτε ότι κάτι θα κάνετε για προστασία των δεδομένων και για τα ε, στάνταρ των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα είπατε αυτά, αλλά θέλω να ξέρω κυρίως εσείς τι θα κάνετε για αυτήν την ανισορροπία ισχύω. Ε, θα, θα αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο, ε, θα σταματήσετε αυτό το micro-targeting, αυτή την μικροστόχευση, θα την απογορεύσετε τελείως. Βεστάγερ. Ένα από αυτά που έμαθα από τον καπιταλισμό της επιτήρησης είναι το ότι δεν κάνουμε αναζήτηση με το Google. Το Google μας αναζητά και μας ψάχνει. Άρα το θέμα είναι ότι ξέρουν όχι μόνο τι θέλουμε να αγοράσουμε, αλλά και τι σκεφτόμαστε. Άρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Και συμφωνώ 100% με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Πρέπει να σπεύσουμε. Και είναι πολύ καλή αρχή ο κώδικας διοντολογίας για να προχωρήσουμε σωστά. Γιατί δεν θα πρέπει να μην θυγούν οι εκλογές μέσω της νομοθεσίας. Επομένως, να έχουμε αυτό σαν σωστή αφετηρία. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το νομοθέτημα για τις ε, ψηφιακές ε, υπηρεσίες δεν ξέρω τι θα γίνεται στις λεπτομέρειες η ρύθμιση, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το GDPR, τα δικαιώματα δηλαδή των πολιτών, οι εθνικέ αρχές, θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουν την νομοθεσία και θα πρέπει να ανταποκριθεί και η αγορά και να έχουμε προστασία του ιδιωτικού βίου, να είναι πραγματική επιλογή αυτή και τελικά να έχουμε Δείτε τι αντίδραση στην αγορά και έτσι με έναν καινούριο τρόπο να υπάρχει το περιθώριο κάποιος να βλέπει κριτικά όταν του ζητούν να σε μια αποδοχή όρων. Και λόγω του, του, του, έργου του Κοινοβουλίου τώρα επιβάλλεται ε, η σχετική νομοθεσία προστασία του καταναλωτή. Αλλιώ ε, είναι κάτι αυτό κάτι που φοβίζει. Να μπορεί κανεί δηλαδή να έχει το περιθώριο να πει όχι. Ναι, να έχουμε νομοθεσία. Αλλά και ο πολίτης να ξέρει τι στυλ ζωής θέλει να επιλέξει, δημοκρατία και έχετε κάποια επερώτηση ακριβώς για το θέμα ε, της δικαιοσύνης ε, και της εμπιστοσύνης. Ακούσαμε για την ε, αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά υπάρχει και κίνδυνος δυσμένους διάκρισης. Γυναίκες, έγχρωμοι, λοάδικοι πολλές φορές από τα σχετικά συστήματα της συντηρητικής νομοσύνης αδικούνται. Και στο πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών η Επιτροπή, τι θα κάνει ούτω ώστε αυτά τα συστήματα συνολικά να μην οδηγούν σε δεσμενεί διακρίσεις, κυρίω όσον αφορά αυτού του ανθρώπους. Απάντηση. Ναι και εγώ προβληματίζομαι όντω. θέλουμε να υπάρχει ε, ισότητα ανδρών και γυναικών στην κοινωνία. Μα η τεχνητή νοημοσύνη κάνει ό,τι της λες, ό,τι δεδομένα της δίνεις. Άρα, εκεί είναι το κλειδί. Ο άνθρωπος το κανονίζει το πλαίσιο και ο κίνδυνος είναι αν κανείς δεν κάνει τίποτα, τότε παγιώνονται αυτές οι προϋπάρχουσες ανισότητες. Αντί να κάνουμε ό,τι πρέπει από το χέρι μας για να αλλάξει κατάσταση και μία από τις αρχές του να είναι ε, αξιόπιστη την την νοημοσύνη είναι αυτό, ότι θα πρέπει κάποιος να σχεδιάσει την νοημοσύνη ή να υπάρχει συνεχής εποπτεία από ανθρώπους για συνεχείς διορθώσεις. Πολύ σημαντικό. Και βλέπουμε ποια είναι η αντίδραση από τις επιχειρήσεις για όλες αυτές τις ε, αρχές καθεντήριες που είπαμε και το θέμα είναι πώς θα κοπεί η δυσμενής διάκριση και αυτό είναι πολύ θεμελιώδες στο σε τι πλαίσιο θα κινηθούμε, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη στην τεχνολογία. Πρόεδρος, Αλεσάνδρα Μπάσου, ΙΜΚΟ, ID. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχετε δηλώσει πολλές φορές ε, πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και σκοπεύετε να εργαστείτε για να αναπτύξετε τα κατάλληλα μέσα για να υπάρχει αυτός ο ισότιμος ανταγωνισμός και στην εσωτερική αγορά και ιδιαίτερα στο παγκόσμιο επίπεδο. Ο στόχος αυτός μου φαίνεται κάπως φιλόδοξος να πω την αλήθεια δεδομένου του ότι ξέροντας και την ε, χώρα μου δεν ε, καταφέραμε να το κάνουμε σε μια κατάσταση πολύ πιο απλή όπως στην περίπτωση Τέρκας όπου ε, προκάλεσε, όπως ίσως ξέρετε, την κατάρρευση τεσσάρων ε, τραπεζών και έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση καταθέτες και καταναλωτές. Αναρωτιέμαι λοιπόν ποια θα είναι τα μέσα που θα αναπτύξετε για να εγγυηθείτε τον ανταγωνισμό στο παγκόσμιο ε, επίπεδο για να μπορέσει η Ευρώπη να παίξει επίση όρις. Ακριβώς ε, ο τομέας ε, των τραπεζών είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει υποφέρει πιο πολύ από την οικονομική κρίση και τώρα που έχουμε ανάπτυξη στις χώρες ε, της Ευρωζώνης ε, και αλλού. Αλλά ακόμα για πολλές επιχειρήσεις είναι δύσκολο να ξεπληρώσουν τα δάνειά τους και αυτό φαίνεται και στον ε, τραπεζικό κλάδο ότι έχουν δηλαδή μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Γι' αυτό θέλω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να λέμε, λέμε ότι τώρα είναι όλα καλά και επιστροφή στην κανονικότητα κτλ. Κάθε περίπτωση στον τραπεζικό κλάδο είναι διαφορετική. Αυτό το οποίο κάναμε εμείς είναι βεβαίως να διασφαλίσουμε την προστασία των φορολογουμένων και της αξίας στο μέγιστο δυνατό. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι που και που μια τράπεζα θα βγει από την αγορά. Πιθανότητα θα αγοραστεί από άλλη τράπεζα και θα είναι επώδυνο, καμιά φορά πολύ επώδυνο γιατί βεβαίως υπάρχει παραδείγματος χάρη μια παραπλανητική πώληση όπου κάποιοι αγοράζουν ένα προϊόν που θεωρούν ότι είναι απλή αποταμίευση και είναι ασφαλής ακόμα και αν ε, η τράπεζα έχει προβλήματα ενώ στην πραγματικότητα δεν σημαίνει αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κάποια στήματα αποζημίωση σε περίπτωση παραπλανητικών πωλήσεων αυτομάτως εάν ο καταναλωτής είναι σε μια ευάλωτη οικονομική κατάσταση και κατά περίπτωση, στην περίπτωση στην οποία χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να δούμε πόσα χρήματα χάθηκαν. Έχετε και άλλη ερώτηση. Έχω και άλλη μία ερώτηση πάντα στο θέμα του ανταγωνισμού γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι ακριβώς για να μπορούν οι επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν επί ίσης όρης κάτι το οποίο ε, έχει πραγματικά μεγάλη σημασία για να λειτουργεί η εσωτερική αγορά. Οπότε, σας ερωτώ, για να αποφευχθούν περαιτέρω στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά, εάν θα προχωρήσει και αν θα προχωρήσετε και με ποιον τρόπο μια, σε μια αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τον ε, τομέα της ε, ναυτιλίας, ο οποίος ε, δεν περιελήφθη σε αντίθεση με άλλους στο fitness check του Ιανουαρίου που μας πέρασε. Να έχετε δίκιο. Ο κλάδος αυτός δεν περιελήφθη γιατί είχαν μια δική τους διαδικασία, είχαν προχωρήσει πιο μπροστά, υπήρχε μια δημόσια διαβούλευση για να δούμε εάν είναι κατάλληλοι αυτοί οι κανόνες, αλλά είχαν δικούς τους ε, στόχους και έλαβαμε διάφορες απόψεις. Κάποιοι λένε ότι δεν χρειάζονται πλέον, ε, κάποιοι λένε ότι λειτουργεί μια χαρά και κάποιοι λένε ότι πρέπει, ελάχιστοι λένε ότι πρέπει να αλλάξει. Οπότε για τις κατευθυντήριες γραμμές για την ε, ναυτιλία σε μεγάλο βαθμό θα συνεχίσουν ως έχουν. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στον τομέα αυτόν. Ένα από τα πράγματα που επιτρέπουν μια ισχυρή ευρωπαϊκή ναυτιλία είναι το ότι έχουμε φόρο ναζ και ακριβώς προσπαθούμε να ε, εξακολουθήσει να έχει μια νομότητα. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή ναυτιλία και για τις ευρωπαϊκές σημαίες και θα πρέπει ακριβώς να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί όπως πρέπει για την ναυτιλία. Αλλά είχαμε διάφορες περιπτώσεις όπου είδαμε ότι ο φόρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για διάφορους ε, στόχους και έπρεπε να το περιορίσουμε. Οπότε ε, προφανώς θα παραμείνει η προτεραιότητά μας η ναυτιλία. Σας ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Έπινγκ από το ECR και την Επιτροπή Οικονομικών. Κυρία, Προ... Κυρία Επιτροπέ. Έχετε δύο χαρτοφυλάκια. Εκτελεστική αντιπρόεδρος για την ψηφιακή εποχή και επίτροπος ανταγωνισμού. Θα ήθελα να μάθω πώς θα αποφύγετε πιθανά συγκρουόμουν συμφέροντα γιατί η Επίτροπος Ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι ουδέτερη και να διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη ευημερία των καταναλωτών. Η βιομηχανική στρατηγική, από την άλλη, σκοπεύει να προωθεί συγκεκριμένους κλάδους και εταιρείε καθώς και την στρατηγική αυτονομία. Και σημαίνει μια άλλη προσέγγιση όσον αφορά τη βιομηχανική στρατηγική. Αναγνωρίζεται την ένταση μεταξύ του στόχου του ανταγωνισμού και της βιομηχανικής πολιτικής. Πώς θα τα συμβιβάσετε αυτά. Θα υπάρξει ένα λεγόμενο συνικό τείχος όπου οι δύο πτυχές ε, του χαρτοφυλακίου σας δεν θα έχουν μεταξύ τους επαφή. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που έκανα και εγώ στον εαυτό μου. Μη αλλιώ πώς ε, μπορεί να δεχτεί κανείς μια τέτοια πρόκληση, γιατί η ανεξαρτησία στην επιβολή του νόμου είναι κάτι το αδιαπραγμάτευτο γιατί αφορά βεβαίω τα στοιχεία, τα γεγονότα, την ε, ε, νομολογία, ούτε το από ποια χώρα είσαι, ούτε τι μέγεθος έχεις και τα Δύο διαφορετικές προοπτικές λοιπόν υπάρχουν εδώ πέρα. Το ένα είναι αφενός το ότι Υπάρχει μια διάρθρωση εντό τη ε, Κομισιόν, δηλαδή η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και η Αρμόδια επίτροπο είναι μέλος ε, της Κομισιόν. Και ήταν ε, έτσι από την αρχή. Έτσι λοιπόν ήταν πάντα, δηλαδή η Επίτροπος Ανταγωνισμού ήταν μέλος της Επιτροπής και οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται και στα θέματα του ανταγωνισμού είναι απόφαση ολόκληρη της Επιτροπής. Βεβαίω αυτό δικαιολογείται γιατί κάθε απόφαση ελέγχεται νομικά όχι μόνο μια φορά αλλά και δύο αν χρειαστεί. Και η τελευταία επιβεβαίωση αυτού ήταν δύο αποφάσεις του 2011 όπου εξετάσαμε το εάν το σύστημα αυτό που έχουμε αυτές τις ομόφωνες αποφάσεις και το δικαστήριο που ελέγχει και την ουσία και την ομότητα της υπόθεσης εκ των υστέρων αν ήταν σύμφωνο με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πράγματι ήταν. Οπότε τα πράγματα είναι σωστά έτσι. Το άλλο είναι το πόσο θα λειτουργεί στην, ε, σε καθημερινή βάση. Και βεβαίως ε, κάτι το οποίο με έχει διακρίνει στη δουλειά που κάνω είναι ότι εγώ και οι ομάδες μου λαμβάνουμε τις ανεξάρτητες συμβουλές του επικεφαλής οικονομολόγου μας και της νομικής υπηρεσίας. Και η νομική υπηρεσία γνωρίζει ότι θα πρέπει αυτά να τα υποστηρίξει και στο δικαστήριο, Κατ' το σημαίνει ότι είναι πολύ προσεκτική να μην υπάρχει παρέμβαση σε οτιδήποτε. Και για τον επικεφαλής οικονομολόγο να μας δώσει μια ανεξάρτητη άποψη για το τι κάνουμε. Ακριβώς όπως λέτε για να διαχωριστεί άσκηση πολιτική από την επιβολή του νόμου. Έχετε και άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ έχουν ανεπτυγμένη πολιτική ανταγωνισμού με παρόμοιου στόχους αλλά διαφορετικέ μεθόδου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα διοικητικό σύστημα ενώ στι ΕΠΑ το σύστημα βασίζεται στο ποινικό δίκαιο. Ο έλεγχο των συγχωνεύσεων είναι πιο συγκεντρωτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυστηρού κανόνε για τις κρατικές ενισχύσεις, ενώ δεν έχει τέτοιες διατάξεις ε, το δίκαιο των ΗΠΑ. Θεωρείτε ότι μπορούμε να διδαχτούμε από τις ΗΠΑ σε κάποιους τομείς και αν ναι, πώς. Μαθαίνουμε πολλά κατά περίπτωση. Έχουμε μια σχέση εργασίας. Όταν, ε, παραδείγματος χάρη, ε, μας ε, όταν δίνεται η εκαθάριση για κάποια συγχώνευση, συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς ομολογούς μας ε, για να δούμε, παραδείγματο χάρη, αν χρειάζεται να απολυθεί κάποιο μετοχικό κεφάλαιο για να γίνει κάτι το οποίο θα ικανοποιεί και εμάς και τους Αμερικανούς ομολόγους μας. Οπότε έχουμε μια συνεργασία και διδασκόμαστε το ένα από τον άλλον. Έχουν ένα διαφορετικό σύστημα στη ΣΥΠΑ, αυτό το, το αναγνωρίζω. Αλλά οι βασικές ιδέες είναι οι ίδιες, γιατί και ε, αρχικά μάθαμε πολλά από τη ΣΥΠΑ και όταν μιλάμε για το αντιτράστη, τον έλεγχο των σχονέψεων αυτά τα πήραμε από τις ΙΠΑ αρχικά. Οι κρατικές ενισχύσεις είναι μια ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα, αλλά αυτό το οποίο πρόσεξα είναι ότι υπάρχουν διάφορε φωνές της ΕΠΑ που αρχίζουν να αμφισβητούν π.χ. το ότι μεμονωμένα κράτη-μέλη θα... Ε, με πολιτείες μάλλον τον είπαμε, συγχωρείτε, δίνουν ε, φόρο απαλλαγές σε εταιρείε για να εγκατασταθούν εκεί. Οπότε όλοι όσοι ασχολούνται με τα θέματα του ανταγωνισμού τα συζητάνε για να δούμε το τι θεωρούμε κατάλληλο σε κάθε δικαιοδοσία. Σας ευχαριστώ. Μάρτιν Σίρτεβαν από την Γκουε και την ΙΜΚΟ. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Είπατε πως θέλετε μία δίκαιη κοινωνία. Χαίρομαι για αυτό. Αυτό κάνει και η δική μας πολιτική ομάδα και στο πλαίσιο αυτό ζητάμε και δίκαιη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Είπατε πως είστε υπεύθυνοι για την εισαγωγή ψηφιακής φορολογίας, ε, φορολογίας των ψηφιακών επιχειρήσεων. Το Κοινοβούλιο στην τελευταία θητεία έχει υποβάλει μια πάρα πολύ προοδευτική πρόταση για το τι μορφή θα μπορούσε να έχει μια τέτοια φορολογία, Παραδείγματος χάρη εκεί πέρα που λαμβάνει η χώρα. Η οικονομική δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι και η φορολογία. Θα ε, υποστηρίξετε αυτή την πρόταση στους ε, G20 και αν αποτύχουν εκεί οι διαπραγματεύσεις γιατί είναι αντιφατικά τα συμφέροντα θα επαναφέρετε την πρόταση αυτή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πώς σκοπεύετε να ξεπεράσετε το μπλόκο στο Συμβουλίο. Είναι δύσκολο να είναι κανείς πάντοτε αισιόδοξο ε, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή φορολογία και τη σχετική νομοθεσία, γιατί παίρνει χρόνο και όταν έχουμε αποτελέσματα ε, πάλι παίρνει χρόνο η εφαρμογή επιτόπου. Όμως, παρόλα αυτά, εγώ προσωπικά εξεπλάγει γιατί πράγματι βλέπουμε πρόοδο. Παρόλα αυτά, όταν ήμουν υπουργό ε, στη Δανία και επιδανική ε, Προεδρία, πήγαινα στο ΕΚΟΦΗΝ και πιέζαμε κάποιε από τι φορολογικέ προτάσει. Και τότε ένα από του συναδέλφου μου είπε: Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πάνω από το πτώμα μου. Τώρα Κάποια χρόνια μετά η πρόταση έχει, έχει γίνει δεκτή και ζει ακόμη ο συγκεκριμένος. Επομένως μπορούν να γίνουν θαύματα. Επί Μοσκοβισή πέρασαν στο Συμβούλιο με ομοφωνία μέχρι τώρα 14 νομοθετήματα. Επομένω, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Ποιο είναι το πρόβλημα. Έχουμε κανένα δυο πολύ σημαντικά νομοθετήματα που δεν ενεκρίθησαν. Ένα από αυτά είναι για την ε, ενιαία κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων. Αν αρχίσουμε να μιλάμε για ένα κατώτατο εταιρικό φόρο, αν παίζει με του φορολογικού συντελεστέ, ε, μπορεί να μην σημαίνει τίποτα αυτό ο κατώτατο ε, φόρο. Θέλουμε λοιπόν πρόοδο στον τομέα αυτό. Και ίσω χρειάζεται κάτι άλλο γι' αυτό. Το δεύτερο που λείπει είναι οι δημόσιε εκθέσει αναχώρα, το οποίο λειτουργεί στον χρηματοπιστωτικό κλάδο την τελευταία φορά που κοίταξα, ε, εξακολουθούσε να υπάρχει αυτός ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, άρα δεν είναι και τόσο σε αυτές οι εκθέσεις. Σίγουρα καλό είναι να έχουμε τις εκθέσεις δραστηριοτήτων, ε, την κατάσταση ε, εσόδων, εξόδων, του ισολογισμού. Όλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να τα ζητήσουμε. Και εγώ, πώς να το πω, εξακολουθώ να ευελπιστώ ότι με πολλή δουλειά μπορούμε να καταλήξουμε σε μια παγκόσμια συμφωνία. Και αν δεν το πετύχουμε, φυσικά και θα καταθέσουμε και θα πιέσουμε για μια ευρωπαϊκή λύση. Εγώ θαυμάζω όσα κράτη-μέλη λένε θέλουμε μια παγκόσμια λύση, αλλά αν αυτό δεν γίνει πράξη θα προχωρήσουμε μόνοι μας. Γιατί είμαστε οι υπόλοιπε επιχειρήσεις που πληρώνουν αυτού του φόρου. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, έχω. Έχουν πράγματι ε, μείνει εκρεμή κάποια νομοθετήματα για την εταιρική φορολογία, αλλά υπάρχει και το άρθρο 116 που δεν ε, ε, χρειάζεται ομοφωνία. Έχουμε το country by country, country reporting και μπορεί με πλειοψηφία η σχετική νομοθετική πράξη. Και έχετε τον ε, Ιταλό Τζεντιλόνι. Έχει νομίζω κάνει κάποιες ανάλογες ε, με εσάς δηλώσει πως αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί. Άρα έχετε ήδη δύο. Είστε δύο που μπορείτε να ακολουθήσετε αυτή την κατεύθυνση την νέα επιτροπή. Ναι, πράγματι. μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 116. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Τώρα, υπάρχει εξή διαδικασία. Κάθε κρατός μέλος καλείται να συμμετέχει, όμως το 116 λέει αν ένα ή κάποια κράτη-μέλη έχουν διατάξεις που ε, είναι επιβλαβείς προς τον ανταγωνισμό, μπορεί κανείς να ξεκινήσει διαβουλεύσεις για αλλαγή των διατάξεων αυτών. Και αν δεν πετύχουν αυτές οι διαβουλεύσεις, αυτές οι συνομιλίες, κατατίθενται προτάσεις και οι προτάσεις αυτές ε, αποφασίζονται στο πλαίσιο της ε, κανονικής νομοθετικής διαδικασίας. Εγώ νομίζω ότι πράγματι καλό θα ήταν να το διερευνήσουμε ε, αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είναι δεδομένο ότι θα πετύχει το εγχείρημα, αλλά καλό είναι να εκμεταλλευτούμε τα εργαλεία της συνθήκης και αν χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσουμε πράγματι. Ευχαριστώ και εδώ ολοκληρώνεται ο πρώτος ε, γύρος και περνούμε στο δεύτερο γύρο για τον οποίο θα προεδρεύσει η κυρία Βαλεάνα ε, που ε, δεν θα καταθέσω βέβαια, δεν θα κάνω κάποια ερώτηση απλά θα δώσω το λόγο στους διαφόρους ομιλητές με πρώτο τον Μάρκους Φέρμπερ, Έκον ε, και Έλκα. Να επανέλθω κυρία Βεστάγκερ στο ερώτημα Επινγκ. Δεν μου ήταν αρκετή αυτή η απόφαση η απάντηση και αν είχα αποδοτήσει πριν πέντε χρόνια ε, ως Επίτροπος Ανταγωνισμού μπορεί να μην με είχε ε, δυσαρεστεί απάντησή σας αλλά τώρα θα είστε εκτελεστική αντιπρόεδρος. Δηλαδή έχετε τώρα τρία βασικά χαρτοφυλάκια και τότε είχατε ένα. Έχουμε και τη σύγκρουση συμφερόντων που ε, είναι κάτι τελείως διαφορετικό τα πράγματα σε σχέση με αυτά που περιγράψατε, γιατί ακούγοντά σας ε, μου φάνηκε σαν να μην χρειάζεται καν επίτροπος ανταγωνισμού, γιατί όλα γίνονται ανεξάρτητα στη Γενική Διεύθυνση. Όμως ε, στην Επιτροπή Γιούγκερ στην οποία ανήκετε ή ανήκατε, υπήρχαν σαφείς κανόνες. Το είχε υποσχεθεί ο κύριος Γιούγκερ και στην αρχή της θητείας, ότι οι φάκελοι της δικής σας Γενικής Διεύθυνσης δεν ε, μπορούν να τις ε, επηρεάσουν άλλοι επίτροποι. Τώρα, αυτά τα εγγενή, αυτή την εγγενή σύγκρουση συμφερόντων με τα θέματα του δικού σας χαρτοφυλακή, πώς θα την επιλύσετε. Η απάντηση. Έχετε δίκιο ότι πρέπει να το δούμε με μεγάλη προσοχή. Είχαμε πράγματι ένα διακανονισμό Σίγουρα έχω την ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους μου όταν χρειάζεται να λάβουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Είναι όλο το σώμα των τρόπων που τις παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάποια σε βάθος ε, συζήτηση ό,τι αφορά τις ε, αποφάσεις για τον ανταγωνισμό, αλλά ακολουθούμε τη διαδικασία, όλα τα βήματα, ε, την εβδομαδία συνάντηση του πολιτικού γραφείου, περιφτάσουμε και οι αποφάσεις δηλαδή λαμβάνονται συλλογικά τελικά. Έτσι πρέπει να γίνεται άλλωστε. Το δεύτερο. Ναι, είναι εντυπωσιακό ο τίτλο του χαρτοφυλακίου μου και ο τίτλο και το περιεχόμενο του χαρτοφυλακίου μου είναι εντυπωσιακό. Όμω, οι νομοθετικέ προτάσει ε, θα γίνουν από του συναδέλφου επίση τη ε, ενιαία αγορά, των εσωτερικών υποθέσεων. Δεν θα τα γράφω λέγω. Ναι, θα συνεργαστώ με τους άλλους επιτρόπους. Αλλά σε ό,τι τις μεμονωμένες προτάσεις, αυτές θα προέρχονται από τους συναδέλφους μου. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην υποτιμούμε και αυτό το οποίο λέει συνθήκη για τον τρόπο ε, λειτουργίας ε, της Ένωσης. Έχουμε την αδιαπραγμάτευτη ανεξαρτησία της επιβολής της νομοθεσίας. Και από την άλλη πλευρά τα ωφέλη των γενικότερων ε, πληροφοριών, ε, επιχειρηματικών πληροφοριών. Αν δεν τα έχουμε όλα αυτά, δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Υπάρχει επιβολή της νομοθεσίας και ρύθμιση. αυτά τα δύο κάπως συνδέονται μεταξύ τους. Μιλήσαμε για τις ε, μεγάλες τεχνολογικές εταιρείε, τα δεδομένα, τι θα πει κανείς ουσιαστικά να έχει μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Και βλέπουμε ότι χρειάζεται κάπου ρύθμιση, άρα πρέπει να πάρουμε αυτά τα οποία λέει η συνθήκη, να τα μετρήσουμε. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με τις αποφάσεις του δικαστηρίου δηλαδή σε συνάρτηση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα σε διάφορες αποφάσεις σε ό,τι αφορά τις ε, ψηφιακές αγορές, ε, πράγματα κινούνται πάρα πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από τις διάφορες νομοθετικές διαδικασίες και πόσο να ε, θα πάρει, παράδειγμα, χάρη, ανάλυση μιας σας θες. Μπορεί να πάρει μήνες μέχρι να αποφασίσετε, θα έχει αλλάξει κατάσταση ε, στην πράξη. Για τον ψηφιακό κόσμο, λοιπόν, χρειαζόμαστε γενικώ πιο γρήγορες διαδικασίες και πιο γρήγορη λήψη αποφάσεων. Έξι χρόνια για την Google έχει αλλάξει εντελώς η κατάσταση μέχρι να καταθέσει τις αποφάσεις και να πάρει ε, μέτρα η Γενική Διεύθυνση. Κύριε Βεστάγκερ. Δύο, πτυχέ. δύο πτυχές θα σχολιάσω. Ξέρετε ότι για πρώτη φορά μέσα σε 20 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία για τα ασφαλιστικά μέτρα, τα προσωρινά μέτρα. Περιμένουμε βέβαια ότι θα αμυνθούν οι επιχειρήσεις σε μια τέτοια περίπτωση. Και το δεύτερο, η δεύτερη πτυχή. Τι είδους εργαλεία χρειαζόμαστε. Ας δούμε τι γίνεται στον Ουρβασίλειο ή στις κατοχώρες. Με ποιο τρόπο προσπαθούν να αναδιοργανώσουν την αγορά όταν ε, οι αρχές ανταγωνισμού διαπιστώνουν ότι δεν τηρούνται κανόνες περί δικαίου ανταγωνισμού. Καλό είναι να οργανωθούμε διαφορετικά πριν υπάρξει πρόβλημα, άρα δεν τιμωρούμε, δεν κολλάζουμε κάποιον, προλαμβάνουμε. Βέβαια μπορεί έπειτα για να πει και το δικαστήριο σε σχέση με αυτούς τους κανόνες, αλλά τι βλέπουμε έχουμε ανταγωνισμό εντός των αγορών, αλλά και για ε, τις αγορές. Παραδείγματος χάρη για την αναζήτηση και την Google συγκεκριμένα. Πρέπει να έχουμε κανόνες, παραδείγματο χάρη, για δίκαιο ανταγωνισμό. Δεν είναι βέβαια ε, σίγουρο ότι θα εφαρμόζονται, όπως είδαμε στην περίπτωση Google 1, 2 και 3. Αυτό το οποίο κάνατε ήταν ε, να επιβάλλετε κάποια πρόστιμα στον τομέα του ανταγωνισμού. Επιτυχή συγκεκριμένα μέτρα. Τώρα όμω δεν είστε ανταγωνιστές είστε στην ψηφιακή εποχή και είπατε ότι θέλετε να αποκαταστήσετε τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη. Πάρα πολύ δημοκρατικό ακούγεται αυτό, αλλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Ε, με τις πλατφόρμες τι θα γίνει. Ε, οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες θα έχουν ε, τα δικαιώματά τους. Οι ανήλικοι επίσης θα προστατευτούν από τα ιντερνετικά παιχνίδια, στοιχήματα κλπ. Πώ θα γίνει η επιβολή του νόμου, πώ θα τα κάνετε αυτά που θέλετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κάτι να γίνει. Er να σα πω. θέλουν στο άμεσο μέλλον, όντω να τα πετύχουμε όλα αυτά και ε, φυσικά και πρέπει να ενεργήσουμε ταχαίω. Πάρα πολλοί νιώθουν απογοήτευση ματέωση γιατί όσοι δουλεύουν σε μια ψηφιακή πλατφόρμα ε, εργάζονται υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Ήδη υπάρχει κάποια εξαίρεση από τους κανόνες του ανταγωνισμού και επομένως εκείνοι οι οποίοι εξομοιώνονται ε, σε, με κάποιον αυτοπασχολούμενο, τότε υπόκειται σε άλλους κανόνες. Άρα και για τις πλατφόρμες και αυτό που θυγανά και σε, άλλες, ε, σε άλλα επαγγέλματα, άρα μπορεί να υπάρχει κάποια συμφωνία με την εργοδοσία και δεν θα είναι θέμα εθνική νομοθεσία. Θα είναι πανευρωπαϊκή η ρύθμιση. Γιατί έτσι κι αλλιώ ψηφιακέ πλατφόρμε καλύπτουν περισσότερα κράτη-μέλη, επομένω ε, αντίστοιχη θα πρέπει να είναι και η οργάνωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Να ένα παράδειγμα του τι μπορεί να γίνει. Επίση, από πλευρά περιεχομένου. Υπάρχει το πρόβλημα του παρανόμου περιεχομένου, αυτό είναι πάρα πολύ βλαπτικό. Ε, στρεβλώνεται έτσι η κοινή γνώμη και αυτό είναι πολύ κακό στις εκλογές, άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Μπορεί να φαίνονται κάπως ε, αυστηρά όλα αυτά, αλλά έχουμε ε, τον κώδικα διοντολογίας. Έτσι μπορούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα σε κάποιο είδους παρόχους του software ε, σε κάποιες μεγάλες πλατφόρμες αυτοί έχουν ήδη συμφωνήσει να υπαχθούν σε αυτή τη ρύθμιση. Άρα το επόμενο ερώτημα είναι χρειάζεται νέα παραπάνω νομοθεσία. Τι θα κάνουμε όμως με την νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ανάγεται στο έτος 2000 αυτή η ρύθμιση. Υπερώτηση κυρία Σαλντεμόσα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, όλα αυτά που συζητούμε, αλλά για να δούμε κάτι άλλο. Έχετε, υποθέτω θα εγκριθεί ο ορισμός σας, έχετε μία πενταετία, ο κόσμος, αλλά και οι εργαζόμενοι, τι θα νιώσουν. Θα προετοιμάσετε τον κόσμο για την ψηφιακή εποχή. Θα είναι, θα είναι τα ωφελιστικά. Και αυτό αφορά και τους ερετούς, τους εκλεγμένους, όπως κάποιοι βουλευτές σε εμά απόκειται να αλλάξουμε την ε, νοοτροπία που υπάρχει και να δούμε τι θα γίνει με τη νέα νομοθεσία. Να γίνουν οι μελέτες των επιπτώσεων, να γίνουν οι ακροάσεις και να περάσει μια νομοθεσία και από εδώ και από το Συμβούλιο. Επομένω, αν θέλουμε να είναι απτά τα αποτελέσματα της δουλειάς μας, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι κανόνες θα θεσπιστούν και θα υπάρξει και συνέχεια. Και όμω να συνεχίσετε και εσείς οι ίδια ε, να εμπλέκετε σε αυτή την προσπάθεια και φυσικά για το νομοθετικό έργο είναι πολύ σημαντικό. Πρόεδρος, Λόκεγκαρτ, Ίμκο. Και άλλο ένα ε, Δανό, θα ακούσουμε και άλλο αυτή την ωραία γλώσσα. Και κύριε Βεσταγκέρ, στις ε, απαντήσεις που μας είπατε ότι είναι σημαντική στήλη τη Ευρωπαϊκή οικονομίας η ΜΜΕ και αντιστοιχούν στο 95% των επιχειρήσεων. Για να δούμε. Από πλευράς νομοθεσία. πώς θα βοηθήσουμε τις ε, ΜΜΕ, Πώ, θα έχουν λιγότερους νομοθετικούς φραγμούς. Τι συγκεκριμένα θα κάνετε γι' αυτό, πώς θα τις βοηθήσετε να αναπτύξουν δυνατότητες στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας, κάποια κατόφλια που να τις διευκολύνουν ίσως. Βεσταγέρ. Κυρίως θεωρώ ότι οι επιχειρήσεις έχουν αρκετά προβλήματα, δεν ε, περιμένουν από μας, αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε να αναπτυχθούν ε, περισσότερο. Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, να κάτσουμε να δούμε τι νομοθεσία χρειάζεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί για τις ΜΜΕ νομίζω το Κοινοβούλιο έχει αυτή την νοοτροπία στο νομοθετικό έργο διότι οι ΜΜΕ αποτελούν την πλειοψηφία και μεταξύ άλλων μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημοσίες συμβάσεις, στους διαγωνισμούς, έτσι να νομοθετήσουμε για τις συμβάσεις αυτές και έτσι να είναι όσο γίνεται πιο ωφέλιμη νομοθεσία των ε, προμηθειών και διαγωνισμών. Να, παράδειγμα ήταν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το χρονοδοτικό μέσο για τις ΜΜΕ, το πρόγραμμα το επενδυτικό του κ. Γιούνκερ. Πρόκειψαν 900.000 συμβάσεις για ΜΜΕ να μην υποτιμούμε το θέμα της προσβασιμότητας από πλευράς εξειδικευμένων εργαζομένων που βοηθούν τις ΜΜΕ. Έχει αυτό και σημασία η παιδεία και η κατάρτιση. Αλλά βέβαια για κατάρτιση και παιδεία δεν έχουμε και τόσες αρμοδιότητες ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες σίγουρα θα πρέπει και οι ΜΜΕ να χρησιμοποιούν, να αξιοποιούν αυτές τις δεξιότητες. Επερώτηση. Σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε. Νομίζω ότι αυτά μας λέτε είναι πάρα πολύ αισιόδοξα, υπόσχονται πολλά, αλλά για αυτό το θέμα του πώς θα έχουν λιγότερους φραγμούς οι ΜΜΕ, να σας πω ένα παράδειγμα. Είναι η οδηγία της προσβασιμότητας και ε, έτσι, βοηθήσαμε. Βοηθήσαμε αυτή την οδηγία της ε, μη της μικροεπιχειρήση. Φτιάξαμε ένα πλαίσιο που βοηθάει. Ε, αυτό απέδωσε, τη ωφέλησε. Ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να εμποδίζει τις επιχειρήσεις αυτές. Άρα θα πρέπει και σε άλλους τομείς ε, ψηφιακούς να κάνουμε το ίδιο. Επίτροπος, ναι, ναι. Το θέλω και εγώ να καταφέρω. Απαιτεί σημαντική προσπάθεια. Ήδη στην Δανία ασχολήθηκα με αυτό που λέτε και είναι δύσκολο να μειώσει κανείς την γραφειοκρατία. Την εικαζομένη, την πραγματική, χρειάζεται έλεγχος μεγάλος, ε, πρέπει κανείς να διαπιστώσει τι γίνεται, τι λύσεις ψηφιακές υπάρχουν που μειώνουν την γραφειοκρατία, ροή δεδομένων να γίνει κάπως διαφορετικά. Χρειάζεται επίσης ε, να δούμε πώς θα γίνει ψηφιακά η μερική απασχόληση. αλλά βέβαια να μην βάλουμε πολύ ψηλά τον πύχη. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρχει ο απεσταλμένος των μιμήσεων που θα μας βοηθήσει από αυτόν. Πιλάρ Δελκάσιο Βέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συμφωνώ 100%. Έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία και η πολιτική μας θα συνάδει με την ψηφιακή εποχή. Και προσπαθούμε να έχουμε άρτια προχωρημένα δίκτυα Το δίκαιο του ανταγωνισμού επίσης έχει βοηθήσει μέχρι τώρα αλλά μιλούμε για υποδομές ψηφιακές, αυτά τα ψηφιακά ηλεκτρονικά πορτοφόλια και άλλες εφαρμογές. Είναι πύλες ψηφιακές για ανταγωνισμό, καινοτομία και πρόσβαση στους πελάτες. Για πετε μας, τι θα κάνετε για να μην υπάρχουν τα μποτιλιαρίσματα που υπάρχουν, περιορισμό δηλαδή στην προσβασιμότητα, στη λειτουργικότητα των ε, λειτουργικών συστημάτων και δεδομένων. Κυρία Βεστή. Κυρία Βέστεγκερ. Νομίζω ότι αν δείτε έτσι τους ε, γενικούς αριθμούς είναι έτσι τα πράγματα, αλλά αν κάποιος ζει ε, στην Ήπεθρο, ε, θεωρεί ότι δεν, δεν, λειτουργεί το σύστημα. Υπάρχει ένα ψηφιακό χάσμα που πρέπει να κλείσουμε για να γίνουν και επενδύσεις ε, εκτός από εκεί όπου είναι αποδοτικό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποιος ρυθμιστής και στο θέμα της υποδομής που είναι πάρα πολύ αναγκαίος νομίζω. Λοιπόν, για αυτή την ε, περίπτωση ε, η νομοθεσία θα έρθει προσεχώς νομίζω μέχρι το επόμενο καλοκαίρι και αυτό θα σας επιτρέψει να ξέρετε το πού βρίσκομαι και αν δεν βρίσκομαι κάπου γιατί ε, συμβαίνει αυτό, αλλά να υπάρχει και ένας μηχανισμός επίλυσης ε, διαφορών, δηλαδή αν τα πράγματα δεν λειτουργούν, ο μηχανισμός δεν λειτουργεί, τι θα κάνουμε για να λειτουργήσει. Αυτό λοιπόν συνέβη με τρόπο πολύ συγκρατημένο, αλλά ταυτόχρονα δημιουργήθηκε ένα παρατηρητήριο έτσι ώστε στην ανάγκη να αυξηθούν αυτές οι υποχρεώσεις. Γιατί βεβαίως εάν δεν εφαρμοστούν οι αρχές της αγοράς, ε, τότε προφανώς έχουμε ένα θέμα και στην ε, περίπτωση τέτοιων υποθέσεων είναι ότι όταν κάποιος έχει de facto κυριαρχία στην αγορά δεν λέει θα διασφαλίσω ισοδομισμό, λέει το δικό μου το προϊόν πρώτο. Οπότε γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να εστιάσουμε στο τι θα συμβεί εάν κάποιος έχει κυριαρχία σε μία από αυτές τις αγορές. Και άλλη για την ε, ψηφιακή υποδομή που είναι μια άλλη διάσταση σε σχέση με την φυσική υποδομή. Με πάση περιπτώσει, σε ένα πλαίσιο στο οποίο πλήττεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται μια ευρωπαϊκή βιομηχανική ατζέντα φιλόδοξη με συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμους ημερομηνίε και συγκεκριμένες δράσεις. Όπως έχουμε κάνει για το κλίμα, από την άλλη ε, λαμβάνοντας υπόψη ε, το ότι αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε μεγάλο στην Ευρώπη είναι μικρό διεθνώς, θα πρέπει να εφαρμόσετε μια ε, βιομηχανική πολιτική. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα έπρεπε να προσαρμόσετε την πολιτική του ανταγωνισμού σχετικά. Σας ευχαριστώ κύριε Βεστάκερ. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για την χρήση των κανόνων είναι παραδείγματο χάρη αυτό το οποίο έχουμε για τις ε, συγκεκριμένα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Έχουμε ήδη έναν τέτοιο συνεταιρισμό για τα μικροηλεκτρονικά 40 επιχειρήσεων που θα ε, μας βοηθήσει πάρα πολύ και στην κλιματική αλλαγή γιατί αυτά τα μικροτσίπ θα χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από αυτά τα οποία έχουμε ήδη. Και αυτό μετά θα μας επιτρέψει η διάχυση της γνώσης και θα ξεκλειδώσει και ιδιωτικές επενδύσεις. Για κάθε ένα ευρώ δημοσίων χρημάτων θα επενδυθούν 2-3 ευρώ από ιδιωτικές εταιρείε. Και μέχρι στιγμής έχουμε μάθει αρκετά ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε αυτούς τους κανόνες, αλλά μπορούμε να τους εφαρμόσουμε στην πράξη με τρόπο πιο ευέλικτο. Εδώ λοιπόν έχουμε άλλο ένα τέτοιο παράδειγμα. σε, όχι στην χύψη κλάδο, αλλά εκεί όπου θεωρούμε ότι υπάρχει ένα λάθος, μια δυσλειτουργία της αγοράς. Και εδώ πέρα ακριβώ θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει μια ανταγωνιστική βιομηχανική πολιτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Καϊλή, κατόπιν από τους uh, Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας οι προσδοκίες μας αυξάνονται, οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω, η πρόεδρος χρησιμοποίησε τον όρο τεχνολογική κυριαρχία. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την παγίδα του υπερπροστατευτισμού. Το δεύτερο θέμα αφορά την αμοιβαιότητα. Έχουμε άλλες κρατικές ενισχύσεις όπως στην Κίνα. Τι κανόνες ε, θα μπουν για τον σχεδιασμό και κατόπιν με βάση τον ε, την εμπειρία σας. Δεν θα πρέπει τώρα να ορίσουμε το τι είναι κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην ψηφιακή εποχή για να καλύπτει και την κατοχή δεδομένων ως ε, στοιχείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Βασταγκέρ. Νομίζω ότι είναι κάτι το πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι θα πρέπει να με το τι αποτελεί ισχύς ε, στην αγορά. Ε, δηλαδή λέμε ότι είναι μερίδιο στην αγορά, το πώς λειτουργεί και τα λοιπά, αλλά όταν κάποιος έχει τη δυνατότητα να συλλέξει πολλά δεδομένα, ίσως να μην έχει τεράστιο τζίρο από αυτή την ε, πλευρά της επιχείρησης, μπορεί να το έχει από τη διαφήμιση βεβαίως, οπότε θα πρέπει να δούμε το πώς λειτουργεί αυτό και έχουμε μάθει πολλά από κάποιες από τις περιπτώσεις συγχωνεύσεων που μάθαμε για να δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα δεδομένα ως κάτι το οποίο θα βοηθήσει την καινοτομία αλλά και ως εμπόδιο στην είσοδο άλλων εταιριών γιατί χωρίς τα δεδομένα αυτό δεν γίνεται και αυτό πλέον αποκτά κρίσιμη σημασία όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη γιατί άπαξ και τα έχεις ε, μπορείς να κάνεις ακόμη περισσότερα. Οπότε πρέπει να συζητήσουμε το τι θα κάνουμε με όλα αυτά τα δεδομένα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το κράτος χωρίς ε, να καταλήξω πολύ στην Αγία Γραφή κάπου έχουμε φτάσει να λέμε μακάρι κατέχοντες ε. λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα στην Ευρώπη, αν σκεφτείτε το τι πρόσβαση μπορεί να έχουν οι υπερυπολογιστέ ε, στι επενδυσει 7 ε, 7-8 ε, τέτοιες περιπτώσει που έχουμε παγκοσμία εμβέλεια υποδομέ και αν σκεφτούμε το τι γίνεται με τον Γαλιλαίο και τον Κοπέρνικα και εδώ πέρα έχουμε δεδομένα εξαιρετικής ποιότητα για τον αγρότη για το να καλλιεργεί καλύτερα, αλλά ε, θα το δώσουμε και σε αυτούς οι οποίοι θα μπορούσαν να το πληρώσουν από μόνοι τους. Αυτή είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να γίνει. Για να μην παίρνουν μόνο οι μεγάλοι, αλλά να έχουν και οι μικροί μια ευκαιρία και μια δυνατότητα. Έχετε και άλλη ερώτηση, ναι, ευχαριστώ. Στον, ε, στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείτε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να γίνει παγκοσμίως παίκτη στην ανάπτυξη ε, επιβάλλοντας και ε, κανόνες δεοντολογίας, ε, παραδείγματος χάρη να προστατεύει πολίτες που αποκλείονται από, τους, από τις ασφαλιστικές εταιρείε με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Και πώς θα μπορούμε να αποφύγουμε ένα πλαίσιο άπλουστευτικό που θα αφορά τελείως διαφορετικούς κλάδους όπως η άμυνα ή ο δημιουργικός κλάδος κτλ. Όπως λέτε οι επιστήμονες ε, παλεύουν να βρουν καλά δεδομένα και από την άλλη έχουμε τεχνητή νοημοσύνη ένοπλη. Οπότε, λοιπόν, ε, όπως σας είπα θα ήθελα να σας ρωτήσω δεν γνωρίζουμε τι γίνεται με τα δεδομένα που συλλέγονται από τα μικρόφωνα και τις κάμερες των τηλεφώνων μας όταν δεν χρησιμοποιούμε εφαρμογές. Δεν θα έπρεπε οι πολίτες να έχουν περισσότερες επιλογές και αν μπορείτε να μας πείτε και κάποια πράγματα για το πώς θα αποφύγουμε τον υπερβολικό προστατευτισμό. Ευχαριστώ κύριε Βέστεγκερ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να παίξουν παγκόσμιο ηγετικό ρόλο χωρίς κάποιες δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές και να πούμε ας κάνουμε ό,τι κάνουν και άλλοι. Αν πάνε όλα τα δεδομένα από παντού και ας επενδύσουμε όλα μας τα χρήματα. Θα χάσουμε έτσι. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργείται για να υπηρετήσει τους ανθρώπους. Αυτό είναι άλλου είδους τεχνητή νοημοσύνη. Η ε, τεχνητή νοημοσύνη με κάποιον σκόπο. Και αν δείτε στο τι είναι καλή η Ευρώπη, την υγεία, το περιβάλλον, κινητικότητα, Βλέπετε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Έχουμε πολλά πράγματα λοιπόν που ε, είναι υπέρ μας, αλλά δεν τα βλέπουμε. Πρέπει να τα εκτιμήσουμε και να τα αναπτύξουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και προφανώς πρέπει να το κάνουμε. Και για να γίνει αυτό, ναι, μπορούμε να γίνουμε πρώτοι στον κόσμο, αλλά η εμπιστοσύνη θα φροντίσει και ο κόσμος να αντιληφθεί ότι αυτό είναι υπέρ μου και όχι εναντίον μου. Αυτό είναι και το νόημα της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Σκοτ Κέιτο από τους Πράσινους και την Επιτροπή Οικονομικών. Χαίρομαι που η εκλεγήσα πρόεδρος της Κομισιόν προτείνει μέσα σε 100 μέρες ε, μια νέα πράσινη συμφωνία. Πρέπει οι κανόνες ανταγωνισμού να στηρίξουν τις ε, κλιματικές επενδύσεις και όχι να είναι αντίθετος. Ε, θα πρέπει σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό κλάδο να αναθεωρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές. Πώς θα στηρίξετε την προσαρμογή σε μια κλιματική μετάβαση που λέει και η επιστολή ανάθεση καθηκόντων, Εστερική έλεγχη για τον έλεγχο τη συνέπεια ε, των αποφάσεων με στόχου ε, για απαλλαγή από τον άνθρακα. Θα τα μελετήσετε αυτά. Τι θα γίνει με τι ε, μειώσει θερμοκηπιακών αερίων, θα περιλαμβάνονται στην αναθεώρηση των καθημερινών γραμμών. Υπάρχουν κάποιες και καλυμμένες ενισχύσεις προς τα ορυκτά καύσιμα και τι θα κάνετε με αυτά στον κανονισμό block exceptions θα περιλάβετε αυτά τα και τι θα γίνει, αυτά τα στοιχεία και τι θα γίνει και με τα αεροδρόμια. Ε, yes, you are... Ξεκινήσαμε ένα πρώτο check-up αν θέλετε και ενδεχομένως θα ακολουθήσει και η επανεξέταση πάρα πολλών κατευθυντήριων γραμμών και Κάτι που προηγείται είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, το ETS. Γιατί, Γιατί θέλουμε να είμαστε έτοιμοι όταν ξεκινήσει νέα περίοδος εμπορίας δικαιωμάτων. Αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη. Θα ξεκινήσουν μάλιστα δημόσιες διαβουλεύσεις ε, σχετικά σύντομα. Και ο στόχος μας εδώ βέβαια είναι ώστε να τον λιγότερη κλάδη να αποζημιώνονται για μέσο ή έμεσο κόστος εκπομπών, πώς να το πω, δεν θυμάμαι πώς το λένε, αυτό που πρέπει να αγοράσουν για να μπορούν να εκπέμπουν, αυτό εννοούσα. Και θα το συζητήσουμε αυτό, ξέρετε, γιατί θέλουμε να είναι ως το πιο μικρός ο κατάλογος και θα το δούμε σε συνάρτηση βέβαια και με τον μεθοριακό φόρο άνθρακα, που είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί οι καθημερινέ γραμμέ για το ETS υπάρχουν ακριβώ γιατί υπάρχει το πρόβλημα τη διαρροή άνθρακα, άρα αυτά θα πρέπει να τα δούμε από κοινού. Και πρέπει να κινηθούμε αρκετά γρήγορα. Για το υπόλοιπο τώρα πακέτο, η Πράσινη Συμφωνία σίγουρα θα μας απασχολήσει. Δεν θέλουμε ε, μάλλον δεν δίνουμε εμεί τι κρατικέ ενισχύσει, αλλά τα κράτη-μέλη. Και εμεί τι κάνουμε, ελέγχουμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Και δεν θέλουμε οι κρατικέ αυτέ ενισχύσει να βλάπτουν τον ανταγωνισμό ούτε το εμπόριο. Οι κατευθύνσει γραμμέ για τι κρατικέ ενισχύσει εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο τη Νέα Πράσινη Συμφωνία. Θα προσπρογράψω τα κράτη-μέλη. Για τα αεροδρόμια. ο κανονισμός Block Exceptions ε, περιλαμβάνει πλέον και τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια. Όσο θεωρούν ότι το χρειάζονται τα κρατημέλη και για λόγους ε, συνδεσιμότητας θα παραμείνει εκεί. Θα παραμείνουν και τα αεροδρόμια μέσα σε αυτόν τον κανονισμό μετάβαση στην πράσινη οικονομία απαιτεί δημόσια χρηματοδότηση για τι βιώσιμε δραστηριότητε. Από την αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης όμως ο τραπεζικό τομέας έχει πάρει 650 δι κρατική υποστήριξη σε κάποιες περιπτώσεις Σε αρκετά συζητήσιμες. Θα ολοκληρώσετε την ανακοίνωση του 2013 για να την ε, ευθυγραμμίσετε με τις νέες διατάξεις ώστε να μην δίνονται χρήματα στο πλαίσιο τη Νέα Πράσινη συμφωνία σε χρεοκοπημένα ιδρύματα. Απάντηση. Απάντηση. Δεν ξέρω πώς να το πείτε, τάση να το πείτε, τέλο πάντων βλέπουμε όλο και λιγότερες ε, τράπεζες να μπαίνουν σε περιπέτειες και αυτό είναι κάτι θετικό. Επίσης βλέπουμε και τα κράτη-μέλη να ενδιαφέρονται περισσότερο για κάποια προγράμματα που δεν έχουν κρατικές ενισχύσεις, ε, αλλά επενδύουν κάποιοι αυτά. Και αυτό είναι σημαντικό για να ξεφορτωθούμε κάποια τοξικά, μη σπερτούμενα δάνεια, που ήταν πρόβλημα σε κάποια κρατημέλη αυτή η ανακοίνωση του 13 για τις τράπεζες κάποιες φορές ε, νομίζω ακόμη ε, είναι η το κατάλληλο πλαίσιο και θα δούμε όταν θα τεθεί σε ισχύ πλήρω τραπεζική ένωση αν θα χρειάζεται ή όχι, αλλά δεν θέλω να βιαστώ υπερβολικά. Γιατί καυστερεί να λήξει η χρηματοπιστωτική κλίση για κάποιες κρίσεις για κάποιες περιπτώσεις. Η ουρά είναι μεγάλη του Γαϊδάρου ακόμη. Και σίγουρα και οι επενδύσει ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ε, είναι κάτι θετικό. Υπάρχει αυτό ο μηχανισμό ε, δυνατοτήτων. Με στόχο ακριβώ να επενδύσουν, να επενδύσουν πολλά στι ανανεώσιμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Επόμενο ο κύριο Ζιβά. ID. Ευχαριστώ κύριε Βεστάγκερ να σας συγχαρώ για τη δράση σας ως Επίτροπο την προηγούμενη πεντέτη. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σε σχέση με τις γραπτές σας απαντήσεις, με ε, πεποίθηση, ε, λέτε ότι εμπιστεύεστε την ε, νέα αγορά. Σε ό,τι αφορά όμως την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά δεν είμαστε στην πρώτη γραμμή. Στην οικονομική ιστορία ποτέ δεν κάλυψε το χαμένο έδαφος μια χώρα σε έναν συγκεκριμένο κλάδο παρά μόνο με προστασία μέσω απαιτητικών δεσμολικών και μη εμποδίων. Πώς θα βοηθήσετε την Ευρώπη λοιπόν να χάσει το χαμένο έδαφος στον τομέα το ψηφιακό και τη στέχνη της νεμοθήνης χωρίς να αμφισβητήσετε κάποιες συνθήκες με βάση τον ελεύθερο δόγμα και έχοντας υπόψη ότι ε, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι έχουν ε, περιχαρακώσει τις αγορές τους. Ε, θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Ευχαριστώ. Ένα από τους λόγους για τους οποίους μεγαλώνουν οι επιχείρηση είναι γιατί εμπορεύονται, έχουν συναλλαγές. Και στην περισσότερη πρόκειται για δοκινοτικό εμπόριο. Στα δύο τρίτα του οι συναλλαγές γίνονται μεταξύ κρατών μελών. Για να, χάσουμε, για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, σε πράγματι. το πόσο ψηφιακά ανεπτυγμένη είναι μια χώρα έχει σημασία. Κάποιες είμαστε, κάποιοι, οι πιο προηγμένοι είναι όσο η Νότια Κορέα και η λιγότερο όσο η Ρωσία. Και πρέπει επομένως να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Uh, και υπάρχει ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των uh, περισσότερων κρατών μελών και βέβαια χρειάζονται και επενδύσεις. Δεν νομίζω να εκτιμάμε πάντοτε επαρκώς στην ευρωπαϊκή ισχύ. Είναι τελείως διαφορετικά τα μοτίβα. στον τομέα των επιχειρήσεων. Αν δείτε αυτά τα περιβάλλοντα, business to business, ε, λειτουργούν κάπως διαφορετικά. Και θα πρέπει σίγουρα να τα καλύψουμε όλα αυτά, το ε, υπολογιστική και πολλά άλλα που θα πρέπει να τα χρηματοδοτήσουμε. Άρα βοηθήστε μας να περάσουν ο προϋπολογισμός, να εγκριθεί για να μην χάσουμε χρόνο για τις κρίσιμες επενδύσεις αυτές. Thank you. Follow Ευχαριστούμε. Επερώτηση. Ζουβέν. Ευχαρίστω. Για να διευρύνουμε λίγο την κουβέντα μας. Φοβάμαι ότι πολλές φορές να ξεχάσουμε τι είναι στο παρελθόν και να δούμε τι γίνεται στο μέλλον. Δηλαδή, τι γίνεται με την ε, παρέμβαση της βιομηχανίας και της τεχνολογίας σε φυτά ζώα αλλά και σε άνθρωπο. Ε, ε, νομίζω το κάνουν Κινέζοι και Αμερικάνοι. Ε, βιοτεχνολογία θα είναι ο αγώνας στο μέλλον. Αυτό θα ισχύει σε πάρα πολλά μέτωπα. Εσείς τι προσέγγιστα έχετε σχετικά. Τι σκέφτεστε να κάνετε γι' αυτό. Κυρία Βεστάκη. Θα με βοηθήσει η πιθανός μέλος της συνάδελφης κυρία Γκαμπριέλ, γιατί εκείνη θα αναλάβει ένα γιγαντιαίο ερευνητικό πρόγραμμα του Rise Europe. Αυτό θα είναι μία από τις ε, λύσεις στο πρόβλημα. Θα είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη. Ναι, όπως είπατε, είναι πολυκλαδικό αυτό το μέτωπο, αυτή η προσπάθεια και θα μας βοηθήσει το πρόγραμμα γιατί στο Horizon έχουμε νέα προσέγγιση. ολική προσέγγιση και όχι κατάτμιση της προσπάθειας. Έτσι θεωρούμε ότι θα ανταποκριθούμε σε αυτό το οποίο είναι η πρόκληση και τις εξελίξεις ε, στην επιστημονική κοινότητα. Το Σενόφσκι. ECR για την Ήτρε. Θα σας τα πω στη μητρική μου γλώσσα, πρόεδρε κυρία Βεστάγκερ. Στο κοντινό μέλλον, στα πλαίσια του Horizon 2020, θα επιλεγούν για την τεχνητή νομοσύνη κάποια κέντρα αριστείας. Θα είναι σημαντικό να υπάρξει ισορροπία γεωγραφική. Να εκπροσωπούνται όλες οι χώρες και της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Γνωρίζω τις επιδόσεις ε, της Τσεχίας σε αυτό και θα εκμεταλλευτούν τις δυνατότητε που υπάρχουν, τα περιθώρια επενδύσεων και να ωφεληθούν όλοι, όλη η Ευρώπη. Όλοι να ωφεληθούν όσο γίνεται περισσότερο. Επομένως, να μην επικεντρωθεί η επιτυχία και η ωφέλεια σε συγκεκριμένους τόπους και συγκεκριμένες χώρες. Έτσι θα προχωρήσουμε στην αριστεία και την επιστημονική αριστεία. Δέστε Ναι, και εγώ προβληματίζομαι σχετικά με αυτό. Όλοι να συμμετάσχουν ε, σε αυτή την προσπάθεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχει κάποιο είδου ε, ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων ή μεταξύ διαφόρων τόπων γλώσσες, ε, παραδόσεις, όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν. Και στο Σώμα των Μητρόπων ήδη έχουν πέσει καλές ιδέες. Και να, σας αναφέρω, μία ήταν αυτό το δίκτυο των ε, κόμβων καινοτομίας, και όλα αυτά να μπουν σε ένα κοινό πρόγραμμα, άρα να μην είναι μεμονωμένα το Α ή το Β Πανεπιστήμιο, να συνδυαστούν και προσπάθειε κάποιων προσώπων ε, επιστημονική κοινότητα ε, από διάφορα μέρη της ε, Ένωσης. Φυσικά τα ξέρει καλύτερα κύριε Γκάμπριελ και τώρα κάπως μιλάω εξ ονόματος για λογαριασμό της, αλλά τέλος πάντων η αριστεία θα είναι το κίνητρο, και να τα καταφέρουμε ε, να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Επερώτηση έχετε, κύριε Τωσενόφσκι. ναι, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Πάρα πολύ πιστική. Για πέστε με αυτές τις πρώτες 100 μέρες. Αυτό δεν είναι φιλόδοξο ως ε, προθεσμία στο πρόγραμμά σας. Μας είπατε για μια ευρεία διαβούλευση με αυτό είναι χρονοβόρο, είναι δύσκολο. Ε, μα εν προκειμένου μιλάμε για κάτι πάρα πολύ μεγάλο ως θέμα και σημαντικό για το μέλλον, για την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα πρέπει να έχουμε πολύ γραφειοκρατία, δεν πρέπει να έχουμε νομία. Πού να έρθουν τότε οι επενδύσει. Μήπως ήταν καλύτερα να είναι τα πράγματα πιο απλά και μήπως τελικά δεν αρκούν οι πρώτες 100 μέρες. Ναι, είναι φιλόδοξος στόχος, πολύ φιλόδοξος, οι 100 μέρες και προβληματίζομαι πολύ μεταξύ άλλων για το θέμα που θέλουμε να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη, αλλά θα πρέπει να αφουγκραστούμε ε, τον κόσμο, δεν θα πρέπει να λέμε να κατεβάσαμε μια ιδέα, θα εφαρμοστεί. Θα πρέπει να ακούμε τη γνώμη τι γνώμες μάλλον για την ιδέα. Και να υπάρχει και ισορροπία, μα θέλουμε να προχωρήσουμε σε κάτι καινούργιο, ακριβώ όπω είπατε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην έχουμε πολυνομία. Το ίδιο ισχύει και για τον κανονισμό για τι πλατφόρμες, να νομοθετήσουμε το λιγότερο δυνατόν και κατόπιν να έχουν το παρατηρητήριο ε, και να ξέρουμε τι χρειάζεται και αργότερα να κάνουμε και άλλα στην νομοθεσία. Άρα ε, είναι σημαντικό το feedback από τις επιχειρήσεις που ανέλαβαν να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές, τις κατευθυντήριες για την τεχνητή νοημοσύνη που θα εμπιστευτεί ο κόσμος, αλλά θα πρέπει να αφουγκραστούμε τις γνώμες ταχαίως. Θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο ώστε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Αλλά όντως επήγε το θέμα. Θα πρέπει να χαραχτεί αυτή η στατική για την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόεδρος. Κύριε Κοκαλάρη, για το ΕΛΚ και την ΙΜΚΟ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε. Πραγματικά πρέπει να φύγουν τα εμπόδια για να λειτουργήσει σωστά η ε, εσωτερική αγορά. E οι ενιαίοι κανόνες θα το καταστήσουν πιο εύκολο για τους Ευρωπαίους να ανταποκριθούν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, ειδικά από ΙΠΑ και Κίνα. Έχετε λοιπόν αυτό το νομοθέτημα περί ψηφιακών υπηρεσιών, το οποίο λέτε ότι θα περιέχει κανόνε περιαστική ευθύνη για τι ψηφιακέ πλατφόρμες. Θα προτείνετε νέου κανόνε για την ευθύνη και το ε, καθήκον το οποίο έχουν να ε, υπάρχει και η αναγκαία ελευθερία για την παροχή υπηρεσιών. Θα τροποποιήσετε τους κανόνες ειδοποίησης και καταβάσματος και αν ναι, τι θα κάνετε έτσι ώστε οι νέοι κανόνες οι οποίοι θα προστατεύουν τους καταναλωτές από την εξαπάτηση θα είναι αποτελεσματικοί αλλά και φιλικοί προς τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Βέσταγκερ. Το πρώτο είναι να γίνει ένας απολογισμός. Τι έχουμε ήδη. Γιατί όταν μιλάμε για διάφορα προϊόντα που έχουν ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, ισχύουν ήδη κάποιοι κανόνες. Κανόνες ασφαλείας, ε, πράγματα που φροντίζουν τα πράγματα να μην παίρνουν φωτιά, να μην βγάζουν πράγματα τα οποία ε, βγάζουν αθυμιάσεις κτλ. Ε, θα πρέπει λοιπόν να μην ε, κάνουμε κάτι υπερβολικό και τελικά να πνίξουμε την ε, καινοτομία και την πρωτοβουλία. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, και αυτό θα ήθελα να το συζητήσω μαζί σας, είναι το πώς θα δω τι θα κάνουμε με την οδηγία περί ηλεκτρονικού εμπορίου, που είναι αρκετά παλιά οδηγία, αλλά κάποια από αυτά τα πράγματα Βεβαίω, ε, είναι ζητήματα αρχή, η ελευθερία παροχή υπηρεσιών και ποια ευθύνη έχει κάποιο αν παρέχει μια υπηρεσία στους πελάτες. Μόλι έγινε μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση για την οδηγία περί πνευματικών δικαιωμάτων, ε, αρκετά διχαστική θα έλεγα, και ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Οπότε πρέπει να γίνει ένας απολογισμός πώς δηλαδή θα επιτύχουμε ε, τον στόχο του να έχουμε προϊόντα τα οποία θα εμπιστευόμαστε, θα έχουμε εμπιστοσύνη στην ιδιωτικότητά μας πριν ε, περάσουμε σε κάποια νομοθετήματα για να γνωρίζουμε το τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε. Είναι λοιπόν ε, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και κάποιο περιθώριο για καινοτομία και τα σχετικά. Και αυτή λοιπόν είναι μια δύσκολη ισορροπία. Σας ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Um, I would like to ε, add θα ήθελα να γνωρίζω εάν η νομοθεσία περιψηφιακών υπηρεσιών θα καλύπτει και την τεχνητή νοημοσύνη ή θα είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την τεχνητή νοημοσύνη. Και Δεύτερον, θα είστε έτοιμοι να προετοιμάσετε αυτή την πρόταση ως κανονισμό και όχι ως οδηγία για να υπάρχει εναρμόνιση προς το συμφέρον της ενιαίας αγοράς. Ευχαριστώ. Κυρία Βέστακερ. Ε, για να απαντήσω, απλά δεν, δεν το ξέρω ακόμα. Το ποια θα είναι η καλύτερη μορφή για να επιλεγεί κανονισμός ε, η οδηγία, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ενσωματωμένη σε προϊόντα. Οπότε για τον λόγο αυτό προϊόντα τα οποία, στα οποία είμαστε συνηθισμένοι όπως ένα ψυγείο. Έχουμε ήδη κάποιον κανονισμό για τις απαιτήσει για να είναι ασφαλή. Μετά τι γίνεται αν ενσωματωθεί τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό το ψυγείο για να γεμίζει μόνο του. Και πώς θα φροντίσουμε ότι αυτή η επιλογή είναι η δική σου και όχι κάποιο άλλο. Γι' αυτό ακριβώς όταν μπαίνουμε σε έναν κανονισμό θα φροντίζουμε να γίνεται αυτό επειδή το ε, χρειαζόμαστε. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι να είναι ασφαλείς οι καταναλωτές, να εμπιστεύονται το προϊόν. Να είναι σίγουροι ότι ελέγχουν αυτό το προϊόν. Αυτό θα είναι ο στόχος μας. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα προεδρεύσει η κυρία Ντεσιούτερ της ΙΜΚΟ. Η επόμενη είναι η κυρία Στέφανη κουρτε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε και τις Επίτροπε, σήμερα έχουμε την πράξη δύο βεστάγκερ, ε, όπως ε, ε, τηλεοπτικές σειρές. Ελπίζω να μπορούμε να πούμε, όπως λένε στις διαφημίσεις, ε, σας άρεσε η πρώτη σεζόν, ε, θα λατρέψετε τη δεύτερη σεζόν, Βεστάγκερ. Ιδίως για τα ψηφιακά πώς θα αντιμετωπίσουμε ε, τις μεγάλες αυτές εταιρείες ε, που μετακυλίουν ε, τα πρόστιμα στις, στους και τελικά δεν τους φοβίζουμε και τόσο με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει και η τελική έσχατη λύση που είναι η διάσπαση ή τι θα γίνει για να μπούμε στο top 10 της ψηφιακής οικονομίας, από το οποίο α, ε, είμαστε απόντες στην Ευρώπη. Υποχρεωτική πρόσβαση και διάδοση δεδομένων υπέρ των καταναλωτών και πιο δίκαιο ανταγωνισμό. Είστε υπέρ. Χαίρομαι που μιλήσετε για σειρές. που υπάρχει για σειρές, υπάρχει σεζόν 2 και κάποιοι πηδάνε από το 1 στο 3, για το 2 πάντα είναι το πιο δύσκολο. Η δεύτερη σεζόν, γιατί έχει γύρει προσδοκίες η πρώτη, τέλος πάντων. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ναι, πράγματι τα πρόστιμα δεν κάνουν αυτό που πρέπει, δεν αρκούν. Ήταν κάτι που τιμωρούσε παράνομη δραστηριότητα κατά παρελθόν τα πρόστιμα. Πρέπει να αλλάξουμε όμως για το μέλλον να του πούμε πρέπει να σταματήσετε να κάνετε αυτά που κάνατε και που έχουν το ίδιο αποτέλεσμα την παράνομη συμπεριφορά που είχατε κατά το παρελθόν. Και θα πρέπει να δούμε αν τα ένδικα μέσα ώστε ο ανταγωνισμός στι αγορέ αυτές να βελτιωθεί. Ε, είναι απαραίτητα. Υπόθεση Google. Εμείς ε, στείλαμε επιστολή για τις διαφημίσεις ε, και την τοποθέτηση πρώτον. Και είπαμε ότι αυτό δεν είναι θεμητό, σταμάτησαν να το κάνουν πριν κάνα δύο χρόνια. Δεν έγινε όμως τίποτα για να βελτιωθεί η αγορά. Επομένως πρέπει να έχουμε άλλες λύσεις και προσεγγίσεις. Έχουμε κάποια εργαλεία. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε σε μια τέτοια για παράδειγμα, ότι θα πρέπει να προβεί σε διαφοροποίηση η διάσπαση. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν λιγότερο παρεμβατικές ε, κινήσεις. Φυσικά και θα δω τι μπορούμε να κάνουμε σε περιπτώσει ανταγωνισμού για να στρέψει ο ανταγωνισμός. Και έχουμε και αυτό το νέο φαινόμενο. Ανταγωνισμό για μία αγορά, όχι μόνο εντός μιας αγοράς. Και ποιος κερδίσει ε, στον ανταγωνισμό βάζει και τους κανόνες, de facto. Εμείς όμως θέλουμε δίκαιο ανταγωνισμό. Πώς θα το πετύχουμε αυτό. Έχουμε μια πλατφόρμα που προτείναμε και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και ως ε, αυτοί που επιβάλλουμε την νομοθεσία. Επερώτηση. Έχουμε πολλές προκλήσεις, παγκοσμιοποίηση, κλίμα, κοινωνία κτλ. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν στεγανά στην πολιτική ανταγωνισμού. Πρέπει να συνεργαστείτε με άλλους για την εμπορική, βιομηχανική, ψηφιακή πολιτική, για να είμαστε οι Ευρωπαίοι πρωταγωνιστές. Πριν νομίζω μιλήσατε και για τους αρευτές. Πώς θα βελτιώσετε τη σχετική νομοθεσία για να έχουμε καινοτόμα σχέδια από την ευρωπαϊκή βιομηχανία μέσω αυτών των σημαντικών έργων κοινού ενδιαφέροντος. για να έχουμε σημαντικά ε, προγράμματα και έργα. Ναι, θέλουμε αυτά τα προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος. Πρέπει να προωθήσουμε κανόνες που έχουμε. Μικρο, ηλεκτρονική, έως εσωρευτές. Ε. Θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι και πιο ταχείς για να φέρουμε στην αγορά αυτά τα προϊόντα. Πρόκειται για πολύ πολύπλοκες διεργασίες ε, με τις σωρευτές, Ξεκινάμε από την πρώτη ύλη, πάμε στις κυψέλες, πάμε στις δέσμες και πάμε μέχρι την ανακύκλωση μετά. Ε, δηλαδή καινοτομούμε και ανανεώνουμε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Πολύπλοκη διαδικασία. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο ε, θα βελτιωθούμε. Και εγώ αυτό θέλω. Καλύτερα να χρησιμοποιώ αυτό το εργαλείο παρά να γυρίσω προς τα πίσω και να το αναθεωρήσω γιατί έχουμε και άλλα σημαντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος. Μας περιμένουν για να μπορέσουν να ξεκινήσουν για το top 10 που είπατε. Αν το βλέπατε 10 χρόνια πριν, στην κατάταξη αυτή νομίζω ήταν ε, η Σέλμον, μια Ολλανδική εταιρεία των καυσίμων από την Ευρώπη. Και άλλες ήταν τραπεζικές ή οκτώ καυσίμων. Πού θέλουμε όμως να είμαστε, σε τι κατάλογο. Αν δείτε ποιες είναι οι παγκόσμιες ε, ε, εταιρείε που είναι πρώτες στην κατάταξη για τα θέματα της πράσινης ανάπτυξης, εκεί η Ευρώπη πρωτοστατεί. Αυτό θέλουμε εμείς. Ε, και επειδή υπάρχει αυτή η ζήτηση, δραστηριοποιούνται και σε αυτό τον τομέα οι επιχειρήσεις. Ιδίω ό,τι αφορά τι επιχειρήσει και ιδίω ό,τι αφορά την Πράσινη Συμφωνία, εκεί εμεί εστιάζουμε. Ευχαριστώ. Τέναντ, μη εγγεγραμμένο από την Παίρνετε ο κάθε ε, υποψήφιο επίτροπο ε, ε, μια επιστολή καθηκόντων και σε εσά λέει ότι θα συντονίσετε το έργο για την ψηφιακή φορολογία για να υπάρξει συνένεση σε διεθνέ επίπεδο μέχρι τα τέλη του 2020 ή να προτίσετε ένα δίκαιο ευρωπαϊκό φόρο. Κατά την άποψή μου, οποιασδήποτε απόπειρε επιβολή κάποιου φόρου θα βλάψουν εξορισμού σχεδόν τον ανταγωνισμό και θα πάνε πολλέ θέσει εργασία σε χώρε που δεν θέλουν να επιβάλλουν φόρο στην ψηφιακή οικονομία. Ερωτώ, αυτό ο νέο φόρο τι μορφή θα πάρει. Με το Brexit τι θα γίνει. Θα προσπαθήσετε να πιέσετε το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit να ακολουθήσει γιατί αλλιώς μπορεί να χαθούν θέσει και να πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ή θέλετε, ε, και επίσης τι θέλετε, όλες οι επιχειρήσεις, μόνο οι μεγάλες πολυεθνικές να το κάνουν αυτό. Ευχαριστώ. Απάντηση. Έχουμε μια διαδικασία στο πλαίσιο του ΩΣΑ για να μπορέσει να επιτευχθεί μια παγκόσμια συμφωνία. Κάποιες από τις προτάσεις ακόμα είναι προσχέδια αλλά μελετούν κάτι το οποίο είχε προταθεί εδώ, στην Ευρώπη, με αυτό τον ε, ψηφιακό φόρο που είχε προταθεί. Άλλες προτάσεις πάνε σε άλλη κατεύθυνση. Ποια θα είναι η έκβαση δεν ξέρω. Ελπίζω όμως να εργαστούν τάχιστα. Γιατί αν θέλουμε παγκόσμια συνένεση, χρειαζόμαστε προτάσεις επιτάπτως για να τις συζητήσουμε. Αν βγεις από αυτή τη φορολογική περιοχή, τι πετυχαίνεις, τίποτα. Το θέμα είναι πού δραστηριοποιείσαι, πού γεννάς κέρδος. Εκεί πρέπει να πληρώσεις και τους φόρους, εφόσον συμβάλλεις και στην κοινωνία που σου δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσει την επιχείρησή σου εκεί. Και αυτή είναι μια από τι αρχέ τι οποίε πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε. Αλλιώς, όλο και περισσότερες εταιρείε θα βάλουν την έδρα τους εκεί που δεν χωράνε, αλλά μόνο ένα γραμματοκιβώτιο με ε, τη διεύθυνσή τους χωράει. Ελπίζω να υπάρξει παγκόσμια συνένεση. Ελπίζω λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι και αυτό μέρος αυτής της συνένεσης. Κύριε Τέναντ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εγώ ευχαριστώ το Θεό που φεύγουμε από εδώ μέσα, γιατί όλες αυτές οι ιδέες περί είναι όλα όσα είναι λάθος με την θέλουμε, εμείς θέλαμε μια κοινή αγορά, ελεύθερο εμπόριο και τώρα βλέπουμε φορολογία χωρίς εκπροσώπηση. Αυτό είναι απαράδεκτο και πηγαίνουμε και προς την λογοκρισία. Η διαφορά μεταξύ των Βρετανών και ημών είναι ότι εσείς είστε υπέρ της εναρμόνισης, εμείς υπέρ της κυριαρχίας. Για εμένα το Brexit είναι ένας καλύτερος τρόπος καλύτερης εκπροσώπησης των ανθρώπων και του να έρθει η λήψη των αποφάσεων πιο κοντά στη δημοκρατία. Συνεχίστε, οπωσδήποτε, εμείς ε, θα φύγουμε. Κυρία Φεστάκερ. Δεν ε, συμφωνώ με την άποψή σας, αλλά σας ευχαριστώ που μας εύχεστε καλή επιτυχία. Thank Σε ευχαριστώ. Η κυρία Εύελιν Ρέγνερ, Σοσιαλδημοκράτες ΕΚΟΝ. Επανέρχομαι στην πολιτική ανταγωνισμού. Είπατε ότι σκοπεύετε να αλλάξετε την εφαρμογή αλλά όχι την ρυθμίση. Πώς σκοπεύετε λοιπόν να αλλάξετε την κατάχρηση των ψηφιακών πλατφορμών, ειδικά από τις γιγάντες εταιρείε. Ε, και επίσης σκοπεύετε να κάνετε την απόσπαση εργαζομένων που πάνε σε άλλες χώρες και πληρώνουν εκεί πέρα χαμηλότερες κοινωνικές εισφορές. Υπάρχει λεγόμενη έκπτωση απόσπασης. Θα αντιμετωπίσετε αυτό το νέο πρόβλημα ανταγωνισμού μεταξύ κρατών μελών όπως το κάνατε με τις πρακτικές φορολογικού ντάμπινγκ. Θα χρησιμοποιήσετε την ομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων. Κύριε Βεστάγκερ. Δυστυχώ θεωρώ ότι το θέμα αυτό ακριβώς δείχνει τα όρια της ε, Λειτουργία ε, του δικαίου του ανταγωνισμού και το πώ πρέπει να λειτουργούν σωστά οι αγορέ εργασίας. Γιατί στο παράδειγμα στο οποίο λέτε, όπου δεν καταβάλλονται οι ίδιες ε, ε, εργοδοτικές εισφορέ και ουσιαστικά οι άλλοι φορολογούμενοι επιδοτούν την επιχείρηση, τον εργοδότη, δεν νομίζω ότι μπορεί να λυθεί αυτό με θέμα με, μέσω του δικαίου του ανταγωνισμού. Είναι θέμα Νομοθεσία της αγορά εργασία είτε στο εθνικό είτε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το οποίο εγώ πάντα εκτιμούσα ήταν ε, η φιλοδοξία που είχαμε να λέμε ότι αν ε, δουλεύει κάποιος στο ίδιο μέρος ε, θα πρέπει να έχει και τον ίδιο μισθό για την ίδια δουλειά. Και θα πρέπει ακριβώς να προσπαθήσουμε να εφαρμοστεί αυτή η αρχή. Δεν έχω να πω κάτι τώρα από την σκοπιά του ανταγωνισμού, αλλά ευχαρίστω να το συζητήσω με τους συναδέλφους των οποίων είναι αρμοδιότητα. Σας ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Ναι. Ε, είπατε πριν. Το CBCR και η Ευρωπαϊκή Φορολογική Νομοθεσία ότι δεν είναι χαμένη η υπόθεση. Τι θα κάνετε για να εγκριθεί το CBCR και είστε διατεθειμένοι να περάσουμε σε ε, έναν ελάχιστο ευρωπαϊκό φορολογικό συντελεστή για εταιρείε. Θα πείτε αυτό το οποίο είπατε πριν στους ε, δανούς ε, συναδέλφους μόνο πάνω από το πτώμα μου. κοιτάξτε, δεν ήταν δεν αφορούσε του ε, Δανούς συνάδελφου και ούτε στα Δανέζικα ακούγεται. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε. Από αυτά τα οποία έχω δει στο θέμα της ε, φορολογία είναι ότι ναι, είναι αργή η διαδικασία, αλλά έχουμε πρόοδο. Και ελπίζω από αυτήν την απόφαση για τις κρατικές ενισχύσεις να πάρουν κάποιες κατευθύνσεις στα κράτη-μέλη. Το ίδιο έχουμε κάνει και για την ερμηνεία των ενισχύσεων και για να προωθήσουμε ακριβώ ε, στην αντίληψη των φορολογικών διοικήσεων του πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε υπάρχει, αν θέλετε, κάποια κατεύθυνση, αν και δεν έχουν αποφασίσει τα δικαστήρια. Αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει έτσι φορολογική δικαιοσύνη. Μόνο ομοθεσία μπορεί να το κάνει αυτό. Ένα συνδυασμός λοιπόν αυτών των πραγμάτων και οι αναφορές ανά χώρα και δεύτερος, δεύτερον ναι, υπάρχει και μια κοινή φορολογική βάση για να μην ε, εκμεταλλεύεται κανείς τις ε, διαφορές. Γιατί βεβαίως έτσι οι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές μετά δεν θα έχουν κάποιο νόημα. Οπότε χρειαζόμαστε όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό. Σας ευχαριστώ η κυρία Νίμπλερ από το ΕΛΚ. Σα ευχαριστώ. Κυρία Βεστάγκερ, αναφερθήκατε στη μεταρρύθμιση του δικαίου της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και ξέρετε πως μας έχει απασχολήσει επί σειρά ετών. Και βεβαίως ε, είναι ένα πολύ επίμαχο θέμα. Η πρώτη μου ερώτηση είναι προσωπικά τι άποψη έχετε για το θέμα αυτό, για τη μεταρρύθμιση αυτή την οποία ανέκρινε το Κοινοβούλιο. Δεύτερον, θα φροντίσετε η οδηγία αυτή να μην νερώσει στην εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Και τρίτον, τι αντίκτυπο θα έχει στην ε, νομοθεσία περί ψηφιακών ε, υπηρεσιών, καθώς ε, είναι και αυτός το τομέας αρμοδιότητός σας. Στον συντονισμό, λοιπόν, ποιος θα πρέπει να έχει την ευθύνη της ρύθμισης αυτών των ζητημάτων. Σας ευχαριστώ, κύριε Βεστάγκερ. Όπως ξέρετε, δεν ήταν άμεση ευθύνη μου, αλλά παρακολούθησα την συζήτηση. Ήταν μια συζήτηση και έντονη και διχαστική, γιατί έδειξε ακριβώς το πώς πρέπει να επιτύχουμε μια δύσκολη ισορροπία. Ειδικά όταν πλησιάζει στο ποιοι είμαστε, τι μπορούμε να πούμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Προσωπικά είμαι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό τώρα να μπορούμε να πούμε ότι θα αποζημιώνονται ε, οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων. Ε, υπάρχει μια τεράστια δυσκολία βεβαίως ε, και δεν νομίζω ότι κανείς από μας θέλει να στερηθεί τα όσα κάνουν τραγουδιστές, ηθοποιοί, συγγραφής ε, κτλ. Οπότε χαίρομαι που πετύχαμε κάποιον συμβιβασμό και βεβαίως τώρα η επόμενη επιτροπή θα πρέπει να δώσει κάποια καθοδήγηση για την εθνική εφαρμογή. Ε, υπάρχει μια συνοχή παρά το ότι τώρα υπάρχει μια κοινή νομοθεσία. Και βεβαίω αυτό θα είναι δύσκολο για την επόμενη Κομισιόν γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό κάποιες από τις συζητήσεις αυτές ε, που είχαν κλείσει με τον συμβασμό να ξανανοίξουν. Νομίζω ότι τώρα το ζήτημα της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας έχει λήξει και δεν πρέπει να ξανανοίξει στο θέμα αυτό της νομοθεσίας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί άμα είναι έτσι θα χάσουμε πάλι κάποια από την δυναμική που είχαμε για την αποζημίωση των κατόχων του copyright. Σας ευχαριστώ άλλη μια ερώτηση για την μετάδοση στο διαδίκτυο αθλητικών γεγονότων. Η Κομισιόν έχει κάνει ήδη μια σχετική δήλωση. Το ερώτημά μου προς εσάς είναι το εξής. Θα ακολουθήσετε αυτήν την δήλωση. Και θα ασχοληθείτε με το ζήτημα τι σκοπεύετε να κάνετε με το παράνομο streaming, την παράνομη μετάδοση τέτοιων αθλητικών γεγονότων. Και νόμιζα ότι είχα προετοιμαστεί, ξέρετε, αλλά με πιάσατε απροετοίμαστη σε αυτό το ερώτημα. Θα είναι δύσκολο και αναγνωρίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα αυτό γιατί τόσα πολλά χρήματα ε, πληρώνει κάποιος για τα δικαιώματα και δεν θέλει να υπάρχει παράλληλα live streaming παράνομο, γιατί αυτό ουσιαστικά βλάπτει αυτόν που έχει επενδύσει για να πάρει τα ραδιοτηλεπτικά δικαιώματα. Όμως θα πρέπει να επανέλθω σε αυτό, γιατί δεν γνωρίζω να σας πω κάτι περισσότερο. Thank you. Next speaker, Madame Cornelia. Η, ε, επομένη, κύριε Κορνίλια ναι, κυρία Βέσταγερ, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω εδώ. Εδώ πίσω είμαι. Στις ε, απαντήσεις σας μιλήσατε πολύ για τον ανταγωνισμό, πόσο απαραίτητο εργαλείο είναι για τη διατήρηση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έτσι τα βλέπουμε και εμείς τα πράγματα όμως. Υπάρχουν περιφέρειες που δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικές και στη Γερμανία Έρχομαι από μια τέτοια περιφέρεια που είμαστε από διαρθρωτικής πλευράς πάρα πολύ ε, αδύναμοι. Έχουμε επίσης προβλήματα σε κάποιες περιοχές ε, που έχουν ανθρακοριχεία γιατί θέλουμε να οδηγηθούμε σε απαλλαγή από τον άνθρακα. Τι θα γίνει λοιπόν με τον ανταγωνισμό όπως είπατε και εσείς ε, θέλετε να υπάρχει ανταγωνισμός και ο ελεύθερος δίκαιος ανταγωνισμός τι ρόλο ε, έχει ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν δεόντως και αυτές οι περιοχές για να μην έρθουν ε, μόνο λύκοι και άλλα ζώα να κατοικούν εκεί, αλλά παραμείνουν και άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές. Ε, τι ενισχύσεις μπορούν να υπάρξουν εκεί, πώς μπορείτε λοιπόν να τα ισοσταθμίσετε αυτά, δηλαδή κάποιες ενισχύσεις από τη μία και ως ελεύθερος δαυσός από την άλλη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βεστάκερ. Ναι. Ο ανταγωνισμό, το είπατε και εσεί, είναι μέρο τη απάντηση. Αναγνωρίζω όμω ότι έχει περιορισμού ε, και όταν έχουμε μια ολόκληρη περιοχή ε, περιφέρεια σε μετάβαση, πρέπει να γίνουν επενδύσει πρώτα και πάνω απ' όλα στον άνθρωπο για να μπορέσουν ε, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη νέα οικονομία που θα προκύψει σε εκείνη την περιοχή. Έχουμε το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Το θεωρώ πολύ καλό εργαλείο και επίση πολύ καλά δουλεύουν και τα κράτη-μέλη. Ε, Παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά τι ενισχύσει που δίνουν ε, σε περιοχέ που εξαρτώνται από τα ανθρακοριχεία ε, για να μπορέσουν να κλείσουν και ο κόσμος να δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις, να βρει νέες δουλειές σε άλλους και σε ό,τι αφορά τη βοήθεια που δίνουμε. Αν υπάρχει κίνδυνος μια εταιρεία να μετεγκατασταθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει αυτό, άρα γιατί να μην δώσουμε σε αυτές τις περιοχές ε, βοήθεια για να παραμείνει μια ε, εταιρεία και να επανέλθει ο ανταγωνισμός που θέλουμε, όμως για να γίνει αυτό πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να μπορεί ο κόσμος να ζει εκεί αξιοπρεπώς. Αν δεν υπάρχουν δουλειές, αν υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες, ε, συγκοινωνίες, ε, πώς θα προκύψει αυτή η νέα εξέλιξη, πώς θα υπάρξει ανάπτυξη εκ νέου. Περιφερειακές αρχές, τα κράτη-μέλη και των πολιτών πρέπει να βοηθηθούν ε, και να αξιοποιήσουν τη βοήθεια κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο βέβαια. Ευχαριστώ πολύ για την επερώτηση. Ε, σε αυτές ε, τις περιοχές που έχουν πρόβλημα ε, δομικό. Είπατε θέλουμε Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική. Ωραία όλα αυτά. Τι όμως πρέπει να κάνουμε διαφορετικά, είπατε κάποια. Αλλά αυτό δεν ήταν μια στρατηγική, αλλά ήταν κάποιες μεμονωμένες προτάσεις κάποια λιθάρα και συγκεκριμένα, αλλά ευρωπαϊκή στρατηγική συνολικά τι ε, μπορούμε να προτείνουμε ώστε αυτές οι περιοχές με τα μέσα που μέχρι τώρα ε, διαθέταμε δεν μπορούσαμε να τις ενισχύσουμε παρά σε, εν μέρη, περιορισμένα. Ε, νομίζω καλό είναι να μιλάμε για μια νέα στρατηγική, αλλά συγκεκριμένα. Τι θα περιλαμβάνει, ποια είναι τα βασικά στοιχεία μιας νέας στρατηγικής, κύριε Βέσταγκερ. Ναι, με συγχωρείτε που δεν ήμουν ε, συγκεκριμένη, το αναγνωρίζω. Και έχετε δίκιο που λέτε ότι δεν ήμουν, γιατί δεν ήμουν πολύ συγκεκριμένη. Λοιπόν, το πρώτο, μια τέτοια στρατηγική δεν θα πρέπει να είναι μόνο για τι μεγάλε επιχειρήσει, γιατί δεν αποτελείται μόνο από τέτοιε η Ευρώπη. Υπάρχουν πάρα πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στον τομέα τη βιομηχανία, ε, που έχουν υπεργολάβου, πάνω από έναν μάλιστα. Εξού και η σημασία του μηχανικού ιστού Πρέπει να καλύψουμε λοιπόν όλες τις ε, βιομηχανίες. Δεύτερο, πρέπει να ενταχθούν ε, τα, όλα αυτά στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Δεν μπορούμε να έχουμε μια βιομηχανική στρατηγική που δεν θα την ενδιαφέρει ο οικολογικός προσανατολισμός ε, και η μετάβαση σε μια ήπειρο ουδέτερη προ τον άνθρακα. Αυτές είναι οι διόψεις του ίδιου νομίσματος. Τέλο. Το θεμέλιο πρέπει να είναι ο δίκαιος ανταγωνισμό. Και δεν θέλουμε να δώσουμε χρήματα μόνο σε κάποιες τομείς ή σε κάποιες εταιρείες ή επιχειρήσεις, αλλά να επενδύσουμε στις αξιακές αλυσίδε, ώστε να μπορέσουν να ευημερίσουν οι διάφοροι τομεί. Ένα καλό παράδειγμα είναι η μακροηλεκτρονική και αυτά τα ευρωπαϊκά project κοινού ενδιαφέροντο. Υπάρχουν κράτη και επιχειρήσεις που ε, συνενώνουν τις δυνάμεις τους ε, για την παραγωγή προϊόντων μικροελεκτρονικής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πάρα πολλούς κλάδους και έτσι βοηθούν να απογευθεί εκ νέου η βιομηχανία μας. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση, Τίμο Βέλκεν, Σοσιαλιστές Δημοκράτες, Γιούρι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπατε ότι αναλαμβάνετε την ψηφιακή ε, εποχή και την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε ένα σωρό προβλήματα όμως και λένε οι επιχειρήσεις ότι θέλουν λιγότερη νομοθεσία ούτως ώστε να υπάρχουν τα περιθώρια για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε όμως το GDPR, έχουμε την οδηγία για την, ηλεκτρονική προστασία του ιδιωτικού βίου, θα πρέπει να παράσχεται εγγύησει για σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπω η προστασία προσωπικών δεδομένων, αποφυγή δεσμένων διακρίσεων ιδιωτικού βίου κλπ. Οπότε θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι χρειάζεται να προστατεύσετε και τον άνθρωπο και να προωθήσετε την εμπιστοσύνη στις νέε τεχνολογίε. Να μην υπονομεύσουμε την ισχύουσα νομοθεσία ή τα ανθρωπινά δικαιώματα θα πρέπει όλα αυτά να τα στρέψουμε εις όφελός μας. Uh, uh, συμφωνώ, συμφωνώ 100% όλα όσα είπατε και στην αρχή και στο τέλος. Αλλά θα τα πετύχουμε όλα αυτά εάν φτιάξουμε την νομοσύνη που την εμπιστευόμαστε. Βάσει βάση των αξιών και έτσι θα υπάρξει εμπιστοσύνη. Αλλιώ η κοινωνία θα την απορρίψει. Δεν θέλουμε, δεν τη χρειαζόμαστε, θα πούνε. Κρίμα θα είναι. Γιατί υπάρχουν δυνατότητε για την ε, μόλυνση αργή του κλίματο, την υγεία, ψηφιακέ τεχνολογίε ε, που ωφελούν πάρα πολύ. Και για αυτό και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι ξεκίνησαμε αυτέ τι κατευθυντήριε γραμμέ για το πώ θα φτιάξουμε την νομοσύνη που να εμπιστευόμαστε. Και αυτέ οι κατευθυντήριε μπήκανε σε κάποιο είδου ε, κριτήρια αξιολογικά και οι επιχειρήσει προσφεύγουν σε αυτέ τι κατευθυντήριε. Άρα δεν ασκήσει επιχάρτου είναι κάτι πραγματικό. Και λένε επιχειρήσει αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε για να αναπτύξουμε τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, λένε. Χρειάζεται νομοθεσία, αλλά τέτοια που να μας δίνει δυνατότητες και όχι να μας τις ψαλίδίζει. Αυτό και για τα δεδομένα, γιατί σεβόμαστε τον άνθρωπο και πέραν των χρηματικών πόρων είναι θέμα του τι κίνητρο υπάρχει, τι στόχους έχουμε και φυσικά όλα αυτά επί τη βάση των αξιών μας. Κύριε Φόλκιν, μάλιστα συμφωνούμε επομένω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την ψηφιακή εποχή το άτομο να μπορεί να αποφασίζει τι θα γίνει με τον ιδιωτικό βίο, να μην είναι απλώ ένα εμπόρευμα ο ιδιωτικό βίο, άρα μια οδηγία και έτσι να υπάρχει ε, κατοχής των αυτών των δικαιωμάτων και με την ε, ε, οδηγία e-privacy θα ληφθεί αυτό υπόψη ότι προβλέπεται από τις επιχειρήσεις δεν θα έχουμε μόνο κριτήριο την αγορά ξεκαθαροί κανόνες και αυτό θα σας ρωτήσω εσείς πώς θα το εξασφαλίσετε ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία για την νομοθεσία των κανονισμών που χρειάζεται για την e και το είπε και για το copyright η κυρία Νίμπλερ. Είπαμε να έχουμε κάποια φίλτρα που θα ανεβάζουμε στο Ιντερνετ και τελικά η ελευθερία του λόγου να μην θίγεται ε, και να γίνει έτσι η εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Φέσταγγε. Ναι, θα χρειαστεί πολλή κουβέντα για αυτό που αναφέρατε στο τέλος θα έχουμε ένα πηγενέλα μεταξύ πρωτεύουσων και ε, επίτροπή και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ομοιογενή εφαρμογή από τα κρατημέλη και να μην έχουμε ε, ανομοιογενή εφαρμογή της ε, οδηγίας ανά κράτο. Μεγάλη προσοχή θα χρειαστεί, διότι ε, συζητήθηκε μεταξύ άλλων ε, αυτό για την ε, θέσπιση της οδηγίας και θα επανέλθουν τα εκείνα τα ζητήματα. Η ελευθερία του λόγου, τα ανθρωπινά δικαιώματα, ε, που θα πρέπει όλα αυτά να τύχουν προστασία και είναι σωστό αυτό. Επομένως αυτά θα συζητηθούν, θα ολοκληρωθεί η συζήτηση και θα επανέλθουν. Πάντοτε χρειάζεται εξισορρόπηση των διαφορετικών στοιχείων. Ναι, γιατί είναι οδηγία ή privacy. Υπάρχουν τώρα κάποια προβλήματα, δεν ξέρω πάντως ε, είναι υψηλής προτεραιότητας και συμφωνώ με σας. Θα είναι σημαντικό βήμα να θεσπιστεί η οδηγία. Δεν πρέπει πάντα να είναι μονοδρομος το να κάνουμε πάσα στο κάθε φυσικό πρόσωπο το ότι θα πρέπει να πάνε να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του γιατί τελικά κουράζουν ε, ε, διάφορες ρυθμίσεις και τελικά κάποιος υπογράφει κάτι και απεμπολεί δικαιώματα. Άρα θα πρέπει με το σωστό τρόπο να προστατευτεί ο καθένας. Στους πράσινους ταμείων Μπουσολάκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βεστάγκερ, εδώ είμαι. Αναφερθήκατε σε θέματα βιομηχανικής πολιτικής ε, και το πώς σχετίζεται με την πολιτική ανταγωνισμού. Είπατε ότι θα αντισταθείτε αν τα κράτη-μέλη θέλουν να νερώσουν τους κανόνες ε, για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων για να δημιουργήσουν μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείε. Εμείς ε, συμφωνούμε. Θα πρέπει να διατηρηθεί ο αποκεντρωμένο δυναμισμό όλων των επιχειρήσεων μικρών και μεγάλων. στι στις γραπτές σας απαντήσεις ε, είδα το τι ακριβώς ε, εννοείται με αυτό το οποίο λέτε να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμό και στην ενιαία αγορά και σε παγκόσμιο επίπεδο και β να επανεξεταστούν οι πρακτικέ πτυχέ επιβολή του νόμου με πτυχέ όπω ο καθορισμό τη αγορά. Οπότε το ερώτημά μου είναι έχετε ε, μεταβάλει άποψη ή μετά από την επανεξέταση του ορισμού θα λάβετε διαφορετική απόφαση σε μια περίπτωση όπως ήταν η Siemens Alstom η συγχώνευση. Ε, εν ολίγης, όχι. Γιατί στην περίπτωση Siemens Alstom το θέμα δεν ήταν τόσο η συγχώνευση. Μιλάμε για δύο μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείε που ήθελαν να συγχωνευτούν αλλά δεν ήθελαν να επιλύσουν τα προβλήματα του ανταγωνισμού που είχαμε ούτε σε μηχανές τρένων, ούτε σε τραμ, ούτε σε σειρμούς μετρό, ούτε σε συστήματα σηματοδότησης, ούτε σε τρένα υψηλής ταχύτητας. Λοιπόν, το ίδιο θα ισχύσει και τώρα. Το θέμα είναι να πούμε το εξής. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει κάπου να στραφεί ο πελάτη, εάν οι δύο επιχειρήσει οι οποίε συγχωνεύονται έχουν υψηλότερε τιμέ και χαμηλότερη ποιότητα. Και να του πούμε ότι ναι, υπάρχει παρόλα αυτά μια αγορά. Καμιά φορά α, αυτό δεν είναι ίσως ο κατάλληλος τρόπος να ερμηνεύσετε την απόφαση αυτή. Και ίσως έτσι να με αντιληφθείτε την αξία των όσων κάνουμε. Είχα δύο πανεπιστημιακού που εξέτασαν ακριβώ 15 υποθέσεις αξιολόγηση τη αγορά και βρήκαν ότι ε, ακολουθούμε λίγο πολύ αυτά τα οποία γίνονται παγκοσμίω. Και έτσι θέλω να ερμηνεύω τους ε, κανόνες μας. Το δεύτερο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε και με άλλους, γιατί η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς προέρχεται από διάφορες πηγές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει πλήρης ε, εφαρμογή και θα πρέπει επίσης να υπάρχει κάποια αμοιβαιότητα. Λοιπόν, προσκαλούν πολλούς ανθρώπους να έρθουν εδώ πέρα και να δραστηριοποιηθούν. Η αγορά των ε, δημοσίων αγορών ε, στην Ευρώπη είναι 14-15% του ΑΕΠ, 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ένα 2 με 12 μηδενικά από πίσω. Είναι πολλά τα λεφτά. Τους ζητάμε λοιπόν, αλλά αυτοί μετά δεν ανοίγουν τι δικέ τους αγορέ. Ε, κοιτάξτε, στο δικό μου το χωριό, αν δεν σε καλούν και εκείνοι, σταματάς και εσύ να του καλείς. Σα ευχαριστώ. Κύριε Μπέζελάγκερ, σας ευχαριστώ και για τις δύο απαντήσεις. Ε, η επόμενη ερώτησή μου αφορά αυτό το οποίο είπατε για την κλιματική αλλαγή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα οποία νομίζω συνδέονται ως ένα βαθμό. Οπότε η ψηφιακή τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει δυνατότητες να γίνουν πιο ουδέτεροι ως προς το κλίμα. Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα, αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας, η βέλτιστη χρήση της ενέργειας μπορεί να μας βοηθήσει να φύγουμε από τις υποδομές τις σχετικές με τα ορυκτά κάψιμα θα κάνετε λοιπόν για να αναπτύξουμε αυτό το θέμα για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και θα προσπαθήσω να περιορίσω την χρήση πρώτων υλών. Σας ευχαριστώ κύριε Βεστάγερ. Κοιτάξτε, ε, ένα είναι προφανώς να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε περισσότερες ψηφιακές ε, τεχνολογίες, γιατί ε, πολλές από αυτές είναι πολύ ενεργοβόρες. Οπότε διάβασα για ένα πείραμα ε, που αφορούσε την κβαντομηχανική, το οποίο όταν ε, πήρε μπρος ο υπολογιστής ε, απορροφούσε ολόκληρη την ενέργεια της πόλης μου. δεν είναι και μεγάλη, αλλά αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που μας απασχολεί είναι ένα πολύ σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και αφορά τις μπαταρίες. Και αυτό το οποίο βρίσκω πολύ ενδιαφέρον είναι να περιληφθούν εδώ πέρα και οι πτυχές της ανακύκλωσης για να δούμε το θέμα των πρώτων υλών, το πώς χρησιμοποιούνται οι μπαταρίες. Να μπει αυτό στο πλαίσιο της ε, καινοτόμου διαδικασίας για να δούμε το πώς θα οργανωθούμε και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την υφιστάμενη νομοθεσία για να αυξήσουμε έτσι την ταχύτητα ε, με την οποία καταπολεμούμε την ε, κλιματική αλλαγή. Και αυτό μπορεί να γίνει ψηφιακά ε, βεβαίω εδώ πέρα μπορούμε να συνεργαστούμε με την κυρία Γκάμπριελ η οποία θα είναι υπεύθυνη για το θέμα αυτό του ορίζοντα τη Ευρώπης και βεβαίω αυτό θα αφορά και κάποιες από αυτέ τι διαδικασίε. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση, κύριο Γκάλαχερ, Renew Econ. Ευχαριστώ. Στη, η επιστολή της Πρόεδρου λέει ότι θα χάξει μια νέα στρατηγία μια ΜΜΕ, της μικρές επιχειρήσεις, τις νεοφυής και θα τους ε, μειώσετε το βάρος από νομοθεσία, τους φραγμούς που υπάρχουν για να προχωρήσουν την ψηφιοποίηση. Άρα το θέμα είναι σε τι περιβάλλον θα κινηθούν στην πράσινη οικονομία, στην ψηφιακή οικονομία, να γίνουν επενδύσεις, έρευνα ε, και ανάπτυξη και να μπορέσουν έτσι να έχουν πιο ευρύς ορίζοντες αλλά και πρόσβαση στις πιστώσεις, στη χρηματοδότηση. Άρα ε, αυτά που κάνατε πριν ως ε, ε, Επιτροπής Ανταγωνισμού και τώρα για τα ψηφιακά είναι τελικά ο στόχος κοινό να κάνετε την Ευρώπη πιο αποτελεσματική. Πώς θα άρετε τους φραγμούς για πρόσβαση χρηματοδότηση για τις μικρές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αναπτυχθούν η κυρία Βέσταγκερ. Έχουμε θεσπίσει νομοθεσία τόσο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια κεφαλαγορά ευρωπαϊκή, αλλά βέβαια άλλο η νομοθεσία και άλλο το να πετυχαίνει κανείς με αυτήν τους στόχους του. Οπότε ε, όλα αυτά ε, ο κύριος Ντομπρόφης τα έχει αναλάβει ε, για την οικονομία υπέρ του κόσμου, για βιώσιμη χρηματοδότηση. Έχουμε τώρα βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτωπο, είναι σημαντικό ε, για την ε, κλασική προσφυγή στην τράπεζα ή την προσφυγή στην αγορά, στην κεφαλαία αγορά, γιατί όταν θέλει κάποιος να ξανοίξει την επιχείρησή του θέλει κεφάλαιο, αλλά θέλει και γνώση από διαφορετικές πηγές που έρχεται πακέτο με το κεφάλαιο, με τα κεφάλαια. Οπότε έτσι γίνεται και έτσι μπορεί μια επιχείρηση να μεγαλώσει. Αυτό είναι ε, μία απόψη της λύσης. Έχουμε όμως τα μέσα για να δώσουμε τη χρηματοδότηση και είχαμε το σχεδίο Juncker που βοήθησε 900.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ε, αυτό είναι παράδειγμα προς και έτσι να δώσουμε τη χρηματοδότηση και να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να μεγαλώσουν. Και ε, μια άλλη πτυχή του θέματος είναι να μπορέσουμε να ε, έχουμε προσλήψεις ανθρώπων κατριτισμένων, με δεξιότητες ευξημένες. Γι' αυτό και έχει σημασία η σοβιακατάρτιση, η παιδεία. Αυτό είναι πια πολύ βασικό εργαλείο, αν θέλει κανείς η οικονομία να προδέψει. Επερώτηση. Ναι. Όσον αφορά τα θέματα των μικρομεσιών, μας είπατε για το upscaling ε, στις επενδύσεις και, και για τους ε, εργαζομένους που καλύτερες δεξιότητες και έτσι κανείς ε, μπορεί να σταθεί δίπλα στις πολυεθνικές. Εσείς τι στρατηγική μπορείτε να έχετε από πλευράς κινήτρων των ΜΜΕ για να επενδύσουν σε αυτά τα μέτωπα όσον αφορά δηλαδή, τους εργαζομένους, κάτι που αναφέρθηκε από πολλούς σήμερα. Επίτροπος, σε συνεργασία τα κάνουμε αυτά με τις εθνικές αρχές, φτιάχνουμε προγράμματα επίσης και έτσι ε, οι εργαζόμενοι αποκτούν δεξιότητες, ε, κατάρτιση, εκμάθηση, εξαποστάσεως. Άλλαξαν τα πράγματα. Δεν έχουμε απλώς παρακολούθηση διαλέξεων από το ίντερνετ. Έχουμε τεστ, παιχνίδια, βίντεο, ε, πληροφορίες, ούτω ώστε έχουμε αυτή την καινούρια μορφή μάθησης και αυτό αποτελεί και πηγή έμπνευσης. οπότε έτσι νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερους και που να αποκτήσουν ψηφιακέ δεξιότητες και αυτό είναι θέμα της κυρίας Γκάβριλ, αλλά όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να τη βοηθήσουμε και έτσι ε, αυτού του είδους η ψηφιακή μόρφωση να προχωρήσει προτεραιότητα. Αλλιώ δεν εκμεταλλευόμαστε τι νοτές που υπάρχουν και το ταλέντο που χρειάζεται. Τελευταία ερώτηση. ίδια Περέρα, ΕΛΚ και Οικονομική Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και κυρία Επίτροπε. Όπως ξέρετε, έχουμε τεράστιες ε, αλλαγές στην κοινωνία από την ψηφιακή τεχνολογία. Κατανάλωση, πληρωμές, ε, ότι αγοράζουμε, θα ε, ε, αλλάξει η ζωή μας και οι εταιρείε αλλά και οι καταναλωτές. βρίσκουν καινούργιες λύσεις από αυτή την τεχνολογία που δεν γνωρίζει σύνορα. Ψηφιακή Ευρώπη ε, αφορά και την ε, φορολογία και το θέμα είναι ότι γίνεται με τι εταιρείε που γεννούν κέρδη σε πολλέ χώρε, τι πληρώνουν σε μία. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει συντονισμό και να δούμε το ότι πρέπει να υπάρξει για ψηφιακή υπηρεσία. Ευρωπαϊκό φόρο και αυτό θέλει και ο κόσμο. Άρα εδώ χρειαζόμαστε συγκεκριμένε λύσει. Εσεί πώ το βλέπετε. Πώ θα γίνει η φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών. κύριε. Ναι, χρειάζεται τέτοιος φόρος. Εδώ αφορά αυτό πολλές επιχειρήσεις, πληρώνουν φόρο, δημιουργούν ε, θέσεις απασχόλησης, προσλαμβάνουν νέους, ε, μαθαίνουν την τεχνολογία, την, την τέχνη και πρέπει να πληρωθεί ο φόρος και ε, πρέπει να εξασφαλιστεί ισονομία και δικαιοσύνη. Και επίσης υπάρχει και ανταγωνισμός σε επίπεδο ψηφιακό για τα, το, το, το κεφάλαιο για τους πελάτες ε, και επομένως δεν είναι σωστό ε, το, το, να μην ρυθμίζεται ο, το θέμα της φορολογίας και θέλουμε να προωθήσουμε ένα τέτοιο φόρο ε, και μετά το κάθε κρατός μέλος θα έχει τη δική του λύση και αυτό το θαυμάζω γιατί είναι πάρα πολύ εξαιρετική ως προσπάθεια και άρα χρειάζεται να ασκηθεί πίεση ούτως ώστε να βρεθεί μια γενική λύση, να υπάρξει γενική συνένεση. Ιδάλλως νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να το κάνουμε. Και βέβαια, αν δεν υπάρξει συμφωνία με το 2020, θα κάνουμε εμείς μια πρόταση. Περέιρα, σε περώτηση. Ναι, για, για ξεκαθαριστή μου όμως. Πώς θα φορολογήσουμε εκείνους που αλλού δημιουργούν τα κέρδη και αλλού είναι εγκατεστημένοι και ε, μεταφέρουν τα κέρδη. Είναι δυνατόν έτσι να φορολογήσετε και έτσι να συρρυκνώσετε τα κέρδη. Προχωράει η Ευρώπη και άρα χρειάζεται μια γενική διεθνής συμφωνία. Δεν θα πρέπει έτσι να περιοριστούν η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και η δυνατότητα έλκυσης επενδύσεων. Τι θα κάνετε, πώς θα λειτουργήσει ο σχετικός φόρος, επίτροπος. Είπα ότι εργάζεται ο ΣΑ επ' αυτού. Την ώρα που μιλάμε, δουλεύουν πάνω σε αυτό. Η πρόταση κατέθεσε ο συνάδελφος Μοσκοβισή ποια ήταν. Μπορείτε να έχετε κέρδος στις συναλλαγές σας με τους χρήστες, μπορείτε να δημιουργείτε όμως αλγορίθμους. Το θέμα είναι πού δημιουργείται η αξία. Είναι εκεί που χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες σας, εκεί που ο κόσμος ε, μένει, μεταφέρεται κτλ. Μπορεί να έχετε σε τελείως διαφορετική χώρα την έδρα σας, αλλά εκεί που χρησιμοποιείτε την υπηρεσία σας από τον κόσμο, εκεί παράγεται και το κέρδος σας. Και παράγεται αξία όταν έχετε συναλλαγές με όλους αυτούς και αλληλεπίδραση με όλους αυτούς τους χρήστες. Και εκεί πρέπει να συμβάλλετε με τα κέρδη σας, δηλαδή να στηρίζετε τη χώρα στην οποία παράγεται το κέρδο σας. Από τότε ε, που ε, εφευρέθηκε η εταιρική φορολογία, πολύ πριν τα ψηφιακά δηλαδή, ε, Το θέμα είναι να καταλαβαίνει η ψηφιακή η εταιρική φορολογία που ζούμε, σε τι κόσμο ζούμε. Γιατί αν δεν ελέγξουμε αυτή την κατάσταση, δεν θα πληρώνει κανείς κανένα φόρο, όσο πιο ψηφιοποιείται η κοινωνία. Δημιουργείται αλυσίδα στην ε, νέα αγορά με έντονο το ψηφιακό στοιχείο προϊόντα που τα ξέραμε θα έχουν ενσωματωμένα ψηφιακά ε, στοιχεία σύντομα και πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Πρόεδρος, ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος γύρος των ερωτήσεων. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη των τεσσάρων επιτροπών που είναι σήμερα εδώ ε, για τις ερωτήσεις. Να ευχαριστήσω την κυρία Βέσταγκερ για τις απαντήσεις. Ε, τώρα ξέρετε κυρία Βέσταγκερ ότι έχετε το πολύ πέντε λεπτά στη διάθεσή σας για να κάνετε μια καταληκτική παρέμβαση. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλύψαμε πολύ ευρύ φάσμα σήμερα. Αν εγκρίνετε τον ορισμό μου, για μένα αυτό είναι η απαρχή μιας σχέσης εργασίας, γιατί δεν πετύχουμε τίποτε αν δεν συνεργαστούμε. Και το δεύτερο είναι ότι όλοι σας έχετε εκλεγεί, έχετε εντολή δημόσια. Εγώ απλά έχω οριστεί. Κάποια κυβέρνηση με επέλεξε και είπε να γίνει επίτροπος. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Διότι μόνο αν εσείς με αποδεχθείτε, είμαι δημοκρατικά, έχω τη δημοκρατική νομιμοποίηση για να κάνω τη δουλειά που με έχει ανατεθεί. Ε, μου σημαίνει, σημαίνει πολλά για μένα λοιπόν, αν επαναλαμβάνω εκλεγώ, να μπορέσω να εργαστώ μαζί σας και να βρω λύσεις σε πολύ δύσκολα ε, ζητήματα. Συζητήσαμε το θέμα των πραγματικών δικαιωμάτων. Θα επανέλθει αυτή η συζήτηση ε, όταν θα χρειαστεί να εφαρμόσουν την νομοθεσία τα κρατημέλη. Ή όταν συζητήσουμε την νομική πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες πάλι θα ξανασυζητήσουμε και τι θα γίνει και με την οδηγία το e-commerce που έχει κλείσει 20 χρόνια περίπου. Πολλά χρόνια για κάτι που έχει να κάνει με ψηφιακή τεχνολογία. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν. Αλλά ας δούμε με τη σειρά τους τα πράγματα. Και λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά αυτό που χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι η χρηματοδότηση. Λεφτά χρειαζόμαστε. Προγράμματα, για να μπορούμε κάτι να κάνουμε. Για να μπορεί ο κόσμος να το δει ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα κονδύλια για να επενδύσουν, για να επενδύσουν στην καινοτομία. Οι ερευνητέ μπορούν να, να χρησιμοποιούν ε, τα κονδύλια για να, δημιουργούν δίκτυα. Ελπίζω λοιπόν να πιέσετε και για το πολιτές μουσουλμικό πλαίσιο. Δεν νομίζω ότι έχουν υπομονή οι Ευρωπαίοι απέναντι σε εμάς. Γιατί υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν πράξη και αυτό πρέπει να γίνει εδώ και τώρα. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω επίσης να με δεχθείτε εκ νέου, γιατί θα ξανάλθω εδώ και θα σας ε, ρωτήσω τη γνώμη σας για κάποια ερωτήματα που δεν έχουμε απαντήσει εκ των προτέρων. Πρέπει να σας συμβουλευτούμε. Το ίδιο θα κάνουμε και με τις ΜΚΟ, την κοινωνία των πολιτών, τους κλάσους βιομηχανίας κτλ. Μιλήσαμε πολύ για τις κατευθυντήριες γραμμές που θα δημιουργήσουν ε, μια τεχνητή νοημοσύνη που θα την εμπιστευόμαστε. Αυτό πώς μεταφράζεται σε κάτι που θα μας δώσει τη δυνατότητα να πετύχουμε τους στόχους μας. Πολύ συζήτηση χωράνε όλα αυτά. Μέχρι να βρεθεί η σωστή λύση. Το σημαντικότερο για μένα και αυτό που θα πάρω μαζί μετά από τη σημερινή ακρόαση είναι το ενδιαφέρον, η προσήλωση, η αφοσίωση σας για τα θέματα που απαρτίζουν το καρτοφυλάκιό Θεμελιώδης αρχές, αξίες, δημοκρατία είναι η βάση μας σε αυτόν τον κόσμο που έχει τόσες προκλήσεις. Με καθησυχάζει το ότι δεν βλέπω κινησμό που δεν λέει κάποιος ας το κάνουμε όπως οι Κινέζοι, αλλά λέμε να το κάνουμε με τον ευρωπαϊκό τρόπο. Εκεί αντλούμε. Ε, από εκεί αντλούμε τη δύναμή μα. Θέλουμε να κάνουμε την Ευρώπη στο δυνατόν καλύτερη για να μπορεί να υπηρετεί όλου μα, όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Και σα ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά. me ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βάσταγκερ, για τις ε, απαντήσεις σας. Δεν ε, μπορώ να προδικάσω το αποτέλεσμα, απλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω αυτή τη στιγμή. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε εδώ πέρα ε, συνάντηση των συντονιστών σε λίγα λεπτά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, λέει η κυρία Τιναγή. Ε, ευχαριστώ εσά, ευχαριστώ κύριε Βεστάγκερ, ευχαριστώ και τι κύριε Βαλεάν και Σούτερ. Ε, σας ευχαριστώ. Λίγα τη συνεδρίαση.